Bene, Ας αρχίσουμε ευθύ αμέσω. Είχαμε βέβαια ένα φορτωμένο πρωινό. Θα συνεχίσουμε όμω στα Ιταλικά. Να πω ευθύ αμέσω ε, ότι έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου παραβίασης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην Ευρώπη. Έχουμε εδώ τους εκπροσώπους του Γραφείου Αναρμόνησης Εσωτερικής Αγοράς ε, και μια ανταλλαγή απόψεων. Το παρατηρητήριο βρίσκεται στο Αλικάντε της Ισπανίας και καλωσορίζουμε τον πρόεδρο του γραφείου, τον κύριο Αντώνιο Καμπίνος, μαζί με τον Δόκτωρ Χόιν. Ε, ο ΕΜΕ, συγγνώμη, είναι η συνδημογραφία του παρατηρητηρίου, δεν είναι όνομα. Ζητά συγγνώμη η πρόεδρος. Και μας ενδιαφέρει φυσικά το θέμα πολύ γιατί όπως ε, είπαν και ορισμένοι συναδέλφοι μας ενδιαφέρει όλο και περισσότερο να καταλάβουμε το έργο σας. Θέλουμε να μαθαίνουμε τα αποτελέσματα των ερευνών και συγκρίσεων που εσείς πραγματοποιείτε σε συντονισμό και με αντίστοιχους εθνικούς οργανισμούς ώστε να μπορέσουμε και εμείς να εξετάσουμε επαρκώς μια πολύ σημαντική προτεραιότητα που θα μας απασχολήσει στους επόμενους μήνες ε, η νομοθεσία περί copyright. Το ζήτημα αυτό της παραποίησης και της πρόληψης της ε, είναι θέμα πολιτισμού. Με πολύ ενδιαφέρον διαβάσαμε μια έρευνά σας ε, ε, για το πώς θα μπορούσαν να ευαισθητοποιηθούν οι νέοι στην Ευρώπη, στα σχολεία της Ευρώπης για το θέμα αυτό αφορά και την ευρωπαϊκή δημιουργική παραγωγή αλλά αφορά και τις μεγάλες επιχειρήσεις που ε, κατέχουν διανοητικά δικαιώματα και συχνά διαμαρτύρονται για την ε, όλο ένα αυξανόμενη πειρατεία, παραποίηση χωρίς επαρκή παρέμβαση. Ο τομέας αυτός αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία σήμερα. Έτσι, σε ένα μήνα, από τις 3 Μαρτίου το 2016, το γραφείο σας θα μετονομαστεί σε Ευρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ένωσης. Η πολιτισμική διάσταση φυσικά δεν μας διαφεύγει. Είναι σημαντική μια ανταλλαγή απόψεων για όλα αυτά και θα θέλαμε να μάθουμε και πώς εσείς αναπτύξατε αυτή την ε, ικανότητα συλλογής και σύγκρισης δεδομένων. Γνωρίζουμε ότι συχνά τα δεδομένα παραποίησης προέρχονται από τις επιχειρήσεις, αλλά δεν είναι απόλυτα βέβαια ούτε συγκρίσιμα. Θέλουμε λοιπόν να μάθουμε πώς προτίθεστε εσείς να συνεχίσετε στο μέλλον της εργασίας σας ε, και τι εργαλεία θεωρείτε ότι υπήρξαν πιο αποτελεσματικά στην πρόληψη και καταστολή τέτοιων τύπων παραποίησης καθώς και τις δραστηριότητες που εσείς έχετε προγραμματίσει. Να δώσουμε λοιπόν αμέσως το λόγο για 10-15 λεπτά στον κύριο Καμπίνος που είναι ο διευθυντής του γραφείου και μετά θα έχουμε μια ανταλλαγή με τους συναδέλφους που θα θελήσουν να κάνουν παρατηρήσεις και ερωτήσεις και μετά θα δώσουμε κάποιο χρόνο για απαντήσεις. Το λόγο έχει ο κύριος Καμπίνο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε αξιότιμα μέλη της Επιτροπής ε, Πολιτισμού και Παιδείας και αγαπητοί βουλευτές. Η ομιλία μου θα διαρκέσει 30 λεπτά. Είχε προετοιμαστεί για 30 λεπτά. Αλλά θα, το κάνω, θα την κάνω συνοπτικά. Λοιπόν, από μνήμης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το παρατηρητήριο παραβέσεις διανοτικών δικαιωμάτων έχει δημιουργηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν δύο χρόνια περίπου βάσει μιας πρότασης ε, της Κομισιόν και μιας ε, συντήφου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το ΟΧΙΜ, για το Γραφείο Εσωτερικής Εναρμόνισης της Εσωτερικής Αγοράς. Όπως θα γνωρίζετε, από τις 23 Μαρτίου θα μετονομαστούμε ε, με την θέση ισχύ του τροποποιημένου ε, κανονισμού για το εμπορικό σήμα για πολλά χρόνια. Στο μέλλον λοιπόν θα ονομαζόμαστε το ε, Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί συγκεντρώνουμε τις αρμοδιότητες που έχει σήμερα το παρατηρητήριο και το γραφείο. Εμείς λοιπόν θα το ονομάζω EUIPO, αν μου το επιτρέπετε, Πού θα είναι η ονομασία αφού τεθεί σε ισχύ ο κανονισμό ένα μήνα. Έχουμε δράσει στο Αλικάντε, απασχολούμε περίπου 2.300 άτομα στα γραφεία μας. Έχουμε ετήσιο προπολογισμό 200 εκατομμυρίων. Έχουμε περίπου 1.300.000 εμπορικά σήματα, σχεδόν 1 εκατομμύριο σχέδια. Βασιζόμαστε απολύτως στο διαδίκτυο. Το 98% των εφαρμογών μας είναι διαδικτυακές. Μόνο το 2% ε, βρίσκεται σε έντυπα. Το ίδιο ισχύει και για σχέδια και για τα σχέδια. Ε, αναπτυχθήκαμε μέσα στην εποχή του διαδικτύου οπότε έχουμε διάφορα εργαλεία πληροφορικής ε, και σε 23 γλώσσες μάλιστα λειτουργούμε σε 23 γλώσσες μπορείτε να βρείτε τα εμπορικά σήματα και τα σχέδια σε 23 γλώσσες και έτσι έχουμε αποκτήσει ειδικευμένες γνώσεις στη διαχείριση και στην ε, εργασία με τα εργαλεία IT. Από τότε που μας ε, δόθηκαν αυτές οι αρμοδιότητες ε, προσπαθήσαμε να ενισχύσουμε το δίκτυο διότι το παρατηρητήριο πρέπει να θεωρηθεί δίκτυο. Δίκτυο όπου συμμετέχουν ιδιώτες και δημόσιοι φορείς. Οι ιδιώτες είναι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, προσπαθούμε να τους πείσουμε να, συμμετέχουν στο παρατηρητήριο και αυτό δεν είναι εύκολο για διάφορους λόγους αλλά προσπαθούμε να προσελκύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και όσοι αποφάσισαν να συνεργαστούν μαζί μας το πράττουν και πολύ επικοδομητικά έχουν τις δικές τους απόψεις αλλά προσπαθούν να είναι επικοδομητικοί και φυσικά έχουμε και εκπροσώπους της βιομηχανίας δεν θα σας εκπλήξει να σας πω ότι έχουμε φυσικά και εκπροσώπους από τα κράτη-μέλη, από το δημόσιο τομέα. Υπάρχει λοιπόν ένα ισχυρό δίκτυο και δραστηριοποιούμαστε και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευρύτερα σε διεθνές επίπεδο ώστε να μπορέσουμε να επεκτείνουμε αυτό το δίκτυο. Διότι ο τομέας της διανοητικής ιδιοκτησίας και της επιβολής του νόμου εκεί ε, χαρακτηρίζονται από πολλούς φορείς, ε, ιδιωτικούς, ε, δημόσιους. Το πρώτο πρέπει να γνωρίζουμε για δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Βρίσκονται εκεί για να αποτελούν ένα μέτρο. Βάσει αυτών βρίσκουμε τις γνώσεις, τις οποίες συνδυάζουμε με τις γνώσεις άλλων, ώστε να εκπονούμε εκθέσεις, μελέτες, βάσει δεδομένων που να μπορούν να έχουν κάποια εφαρμογή, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να κατανοούμε καλύτερα την πραγματικότητα, η οποία ε, είναι δύσκολο. Ε, είναι δύσκολο να έχουμε μια πραγματικά καλή εικόνα της ε, πραγματικής κατάστασης και παρότι έχουν βελτιωθεί τα στοιχεία που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χάρη στο έργο της Eurostat και το Ευρωβαρόμετρο, παραμένει το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές ελλείψεις σε σχέση με αυτό που θα ήταν επιθυμητό ώστε να μπορούμε να δώσουμε στους ε, πολιτικούς, στους εκπροσώπους όπως εδώ των Ευρωπαϊκών Λαών και στα ε, άλλα θεσμικά όργανα ε, να τους παρέχουμε λοιπόν τις σωστές γνώσεις ώστε να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις. Δύο-τρία χρόνια λοιπόν μετά από την μετά από τη μετονομασία του παρατηρητηρίου στο EUIPO ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Ελπίζουμε και ελπίζω να μην σας φανώ αλαζόνας, έχουμε ε, εντονότερη νομιμότητα. Μας θεωρούν έναν ε, νόμιμο δημοσιο οργανισμό, αξιόπιστο, που παρέχει στοιχεία βασισμένα σε ε, μεθόδους διαπιστωμένες, επικυρωμένες, βασίζονται σε μελέτες, με δεδομένα ε, που συνοδεύονται από την εξήγηση από το που προέρχονται και ευρήματα ε, ως αποτέλεσμα των μελετών αυτών. Σήμερα κάποιες μελέτες μας ε, αναφέρονται στους θεσμούς έγγραφα της Κομισιόν, του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου ε, από εταιρείε του τομέα. Έχουμε αναπτύξει ένα σύνολο εργαλείων που θα σα αναφέρω και που χρησιμοποιούν οι βιομηχανίε του τομέα, οι αστυνομικέ αρχέ, ε, οι αρχέ επιβολή του νόμου στι καθημερινέ του δραστηριότητε. Κάποια νούμερα που θεωρώ ότι είναι σημαντικά. Πρώτα απ' όλα, έχουμε κάνει μια μελέτη μετά από μια μελέτη της Αμερικανικής κυβέρνησης βάσει περίπου της ίδιας μεθόδου λοιπόν, που ακολούθησε και η Αμερικανική κυβέρνηση όπου προσπαθήσαμε να δείξουμε σε ποιο βαθμό οι τομείς που χρησιμοποιούν ε, εντατικά την διανοητική ιδιοκτησία Σε ποιο βαθμό λοιπόν οι τομείς αυτοί συμβάλλουν στο Ευρωπαϊκό ΑΕΠ, στην απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο εμπόριο. Και πιστεύω ότι είναι αρκετά εντυπωσιακά τα αποτελέσματα. υπάρχει απευθεία σύνδεση μεταξύ της χρήσης, της εντατικής χρήσης των δικαιωμάτων αυτών και των ε, αριθμών που σας παρουσιάσω. Οι τομείς αυτοί λοιπόν παράγουν αυτό το ΑΕΠ και την απασχόληση που θα σας παρουσιάσω. Αντιστοιχούν κατά 39% σε 40% στο ΑΕΠ. Συμβάλλουν στη δημιουργία 35% άμεσων και έμεσων θέσεων απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τέλος αυτές οι βιομηχανίες, αυτοί οι τομείς ε, συμβάλλουν στο 90%, 90 στο ευρωπαϊκό εξωτερικό εμπόριο. Μια δεύτερη μελέτη που φυσικά μπορείτε εσείς να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΟΧΙΜ ε, που στο μέλλον θα μετανομαστεί σελίδα EUIPO Δηλαδή μπορείτε να πάτε σε αυτή την ιστοσελίδα και να βρείτε τα ευρήματα εσείς οι ίδιοι πέραν των απλών τριών ποσοστών που σας έδωσα διότι η μελέτη αυτή προσπαθεί να δώσει στοιχεία όσον αφορά τις διαφορές μεταξύ διαφόρων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, copyright, σχεδίων κτλ. Ε, και κατά χώρα. Μια δεύτερη μελέτη, επίσης πολύ σημαντική, προσπαθεί να περιγράψει το τι ακριβώς ε, πιστεύουν οι Ευρωπαίοι πολίτες για την πνευματική ιδιοκτησία όπως επίσης και για την καταχρηστική ε, αντιμετώπιση της. Τα ευρήματα δεν εκπλήσουν, τώρα όμως δεν μας εκπλήσουν αλλά ταυτόχρονα τώρα παρουσιάζονται υπό τη μορφή αν θέλετε ε, αποδείξεων. Η μελέτη έγινε σε 23.000 περίπου πολίτες στο σύνολο των κρατών μελών η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν αυτή που χρησιμοποιείται για το ευρωβαρόμετρο. Έγιναν οι σταθμίσεις του ευρωβαρομέτρου. Η μεγάλη πλειοψηφία λοιπόν των πολιτών θεωρεί ότι χωρίς την πνευματική ιδιοκτησία ε, θα βρισκόμασταν σε μια πολύ κακή, ε, θα έλεγα τερματική κατάσταση, θα είχαμε το τέλος του καπιταλισμού να αντιμετωπίσουμε χωρίς την πνευματική ιδιοκτησία, η δημιουργικότητα, η φαντασία ε, θα είχαν σοβαρά προβλήματα. Όταν βλέπει όμως κανείς το τι συμβαίνει στατιστικά και σε εξατομικεύει τις απόψεις αυτές, θα δει ότι το 30% των πολιτών θεωρούν ότι το να αγοράζει κανείς παραχαραγμένα προϊόντα είναι μια μορφή διαμαρτυρίας απέναντι στο καπιταλιστικό καθεστώς, απέναντι στις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Πιστεύουν επίσης ότι σε σχέση με τις παραβιάσεις αυτές κάπου σε ένα βαθμό δικαιολογούνται με λίγα λόγια. Βλέπει λοιπόν κανείς ότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά στην ενημέρωση και τα κενά αυτά είναι πιο σημαντικά ακόμη όταν έχουμε να κάνουμε με πολίτες εκτός αν θέλετε αυτής της αίθουσας 15 με 20 ετών εκεί οι αριθμοί είναι πολύ πιο σημαντικοί των πολιτών δηλαδή που αγοράζουν τέτοιου είδους παραποιημένα προϊόντα και αν συνεχίσουμε λοιπόν στην ίδια πορεία τότε ολοένα περισσότεροι πολίτες θα αμφισβητούν τον ρόλο τον οποίο έχει παίξει στο παρελθόν η πνευματική ιδιοκτησία τα τελευταία 300 χρόνια. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί πέραν αυτών των γενικών μελετών οι οποίες στην ουσία δημιουργούν το πλαίσιο αν θέλετε και θα συνεχίσουμε να τις χρησιμοποιούμε ξεκινήσαμε κάποιες άλλες μελέτες για την παρακολούθηση, την καταμέτρηση της ζημίας η οποία δημιουργείται λόγω ακριβώς της παραβίασης των κανότων των κανόνων της πνευματικής ιδιοκτησίας και της λεγόμενης παρασιτικής οικονομίας. And the numbers here are quite impressive actually. Uh, when, when we look at the five sectors that we've studied, um, Υπάρχουν πολλές μελέτες λοιπόν για κάποια προϊόντα όπως τα κοσμήματα και τα λοιπά και σε άλλους τομείς, για τους πέντε τομείς, η νόμιμη βιομηχανική δραστηριότητα χάνει 55 δις ε, σε σχέση με τον κύκλο εργασιών της. Χρησιμοποίησαμε μία μεθοδολογία που μας δίνει 55 δις. Τα 55 δις σαν δεν λένε ποτέ, 59 δις μάλλον. Εγώ είμαι Πορτογάλος και αυτό σημαίνει το 1 τρίτο περίπου το πορτογαλικού ΑΕΠ, για να καταλάβετε δηλαδή ε, περίπου πώς έχουν τα πράγματα. Κάτι το οποίο είναι πιο σημαντικό, ίσως εξίσου σημαντικό, το οδηγεί σε απώλεια 647.000 θέσεων εργασίας και τα έσοδα των κυβερνήσεων χάνουν περίπου 11,5 δις ευρώ κατέτος, δηλαδή Ίσως αν τα πράγματα συνεχίσουν να χειροτερεύουν τότε θα φτάσουμε στο σύνολο του πορτογαλικού ΑΕΠ και θα προχωρήσουμε και σε ένα μικρό κομμάτι του ισπανικού. Εγώ δεν μπορώ βέβαια να σας δώσω ακριβείς αριθμούς πριν την κυκλοφορία αυτής της σημαντικής μελέτης, αλλά είναι μια μελέτη που κάναμε από κοινού με τον ΩΣΑ Προσπαθήσαμε να καταμετρήσουμε το κόστος των παραβιάσεων αυτών κάτι το οποίο θα δώσει στους πολιτικούς σημαντικά τεκμήρια. Για τις βάσεις δεδομένων τώρα, για μια ακόμη φορά, Προσπαθούμε να προσφέρουμε περισσότερα στοιχεία στη συζήτηση. Έχουμε αναπτύξει μια σημαντική βάση δεδομένων ε, με 280 επιχειρήσεις που μας δίνουν πάρα πολλές πληροφορίες έτσι ώστε να επιτραπεί στις αρχές να διακρίνουν ένα προϊόν για το αν είναι γνήσιο ή παραποιημένο θα υπάρχει και ένα μητρό το οποίο θα επιτρέπει στους υπεύθυνους να γνωρίζουν αν το σήμα του προϊόντος ανήκει στον γνήσιο κατασκευαστή και αν θα πρέπει να δοθεί ή όχι συνέχεια σε μια περίπτωση ή σε μια καταγγελία. Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο, συνδέεται επίσης και με την Τράπεζα Δεδομένων για τα Αντίγραφα που ενημερώνουν τις τελωνιακές αρχές ε, με λειτουργικό τρόπο να καταπολεμήσουν την βιομηχανία των παραποιημένων. Έχουμε και άλλες βάσεις δεδομένων, τις οποίες αναπτύσσουμε με τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης. Έχω 10 λεπτά μόνο και δεν ε, θα ήθελα να ξοδέψω περισσότερο χρόνο μιλώντας για αυτού του είδους τα δεδομένα. ξεπέρασα τα 10 λεπτά. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας, τίποτα άλλο. Thank you. Molto Πολύ ενδιαφέρουσα και ανησυχητική παρουσίαση που κάνατε, τα δεδομένα που μας δώσατε. Δείξατε λοιπόν πόσο μεγάλη ανάγκη έχουμε από το παρατηρητήριό σας και σίγουρα θα υπάρξουν ερωτήσεις από τους συναδέλφους έτσι ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τις εμπειρίες σας και να δούμε ακριβώς τι μαθήματα μπορεί να βγάλει κανείς, τι συμπεράσματα μπορεί να εξάγει κανείς από α, τις εμπειρίες σας και από τους τρόπους που χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση των επιπτώσεων αυτής της παράνομης δραστηριότητας. Η πρώτη συνάδελφος που έχει ζητήσει το λόγο είναι η κυρία Χιμπάτσκα και μετά η κυρία Τρούπελ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ λέει κυρία Λιμπάτσκα. Παρακολούθησα με ζωηρό ενδιαφέρον την παρουσίασή σας. Επιθυμώ να θέσω δύο ζητήματα. Κατά πόσον προτίθεστε να παρακολουθήσετε τις διαπραγματεύσεις για την συμφωνία TTIP διότι είναι πολύ διαφορετικές οι αμερικανικές διατάξεις περί προστασίας της ε, πνευματικής διοκτησίας από αυτές τις ευρωπαϊκές. Δεύτερη ερώτηση. Είπατε και δικαίως ότι οι νέοι 15-20 ετών είναι εκείνοι που παραβιάζουν περισσότερο και συχνότερα το δίκαιο. Γι' αυτό από αυτό απορρέει, απορρέει η ερώτησή μου. Ασχολείστε, προωθείτε σεμινάρια ενημέρωσης των νεαρών αυτών για να αντιληφθούν την αξία της ε, πνευματικής ιδιοκτησίας. Σας ευχαριστώ, η κυρία τρύπελ Σας ευχαριστώ, ε, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για την παρέμβασή σας, κύριε προσκεκλημένη Μιλήσατε για την παράνομη για το παράνομο κατέβασμα περιεχομένου από το διαδίκτυο. Από την άλλη μεριά, εάν έχουμε καλύτερες νομικές υπηρεσίες με καλύτερη ε, προσφορά, θα αλλάξει το σκηνικό αυτό. Ποια είναι η εκτίμησή σας επαρκούν αυτές οι ε, νομικές υπηρεσίες που προσφέρονται ή χρειαζόμαστε και άλλα μέτρα διότι έχουμε μελέτες και αριθμούς που δείχνουν ότι μειώνουν τα μέτρα αυτά ήδη τους αριθμούς των παράνομων ε, του παράνομου downloading. ό,τι αφορά τα εμπορικά σήματα. Πέστε μας λίγο περισσότερο για τη στρατηγική σας. Τι κάνετε για να μειωθεί η παράνομη χρήση. Υπάρχουν άλλα σχόλια ή να κάνουμε ένα πρώτο γύρο απαντήσεων και ενδεχομένω μετά. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Όσον αφορά τις εξουσίες που θα έχετε εσείς, η εργασία σας ε, έγκυται στην παρατήρηση, στη σύγκριση δεδομένων, ευαισθητοποίηση και στο συντονισμό ε, ενδεχομένως θα βλέπετε τα στάνταρ, τα πρότυπα, τους δείκτες που θα προωθείτε με, τους, με τα άλλα παρατηρητήρια, επαλήθευση των αποτελεσμάτων των διαφορών πολιτικών ή και ίσως και αυτός ο προενεργός ρόλος που μόλις είπαμε. Εσείς όλα τα αποτελέσματα σε ποιον τα αναφέρετε, στην Κομισιόν, στο Κοινοβούλιο, έχετε κάποια δυνατότητα να επηρεάσετε και την νομοθετική διαδικασία, τουλάχιστον να σας ακούσουμε, να σας ακούσουν κάποιοι εσάς ως ε, εμπειρογνώμονες στον τομέα. Σκέφτομαι και τη μελλοντική οδηγία για τα πνευματικά δικαιώματα, για το copyright, ε, σας έχει ζητηθεί να παρέχετε πληροφορίες, να συμβάλλετε με κάποιο τρόπο ή δεν είναι αρμοδιότητά σας κάτι τέτοιο. Θα αρχίσω με την ερώτηση της Προέδρου. Λυσμόνησα να σας δώσω σημαντικές πληροφορίες στην πρώτη παρέμβασή μου. Πρώτα-πρώτα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπείται στο παρατηρητήριο στην Ολομέλειά μας εκπροσωπείται και ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας και προσκαλέσαμε 10 ευρωβουλευτές να συμμετέχουν ετησίως στην ετήσια ε, συνάντησή μας. Δεν έχουμε εμείς ούτε νομοθετικές ούτε προνομοθετικές αρμοδιότητες εμείς του παρατηρητηρίου. Μέσω μελετών, ερευνών, συλλέγουμε τα δεδομένα και νομίζουμε ότι μπορούμε έτσι να συμβάλλουμε στην διαμόρφωση πολιτικών. Μπορούμε να συντάξουμε συστάσεις μετά από αίτημα που μας υποβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βέβαια, οι νομοθετικές αρμοδιότητες ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέει ο ομιλητής και βέβαια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτά και σε ό,τι έχει σχέση με την Διατλαντική Συμφωνία. Εκεί βασιζόμαστε στις πληροφορίες που μπορεί να μας δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν παρακολουθούμε ιδιαίτερα την TTIP, αγαπητή κυρία Λιμπάτσκα. Δεν παρακολουθούμε τις διαπραγματεύσεις για την TTIP, παρόλο που Κάθε φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, χρειάζεται κάποια συγκεκριμένη δική μας ε, συμβουλή, την δίνουμε. Έχουμε βεβαίως προγράμματα και δράσεις ε, για να έρθουμε σε επαφή με τους νέους. Έχουμε ένα ταμείο μισού εκατομμυρίου ευρώ για εκστρατείες στο εθνικό επίπεδο αλλά υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με project τα οποία μπορεί να προωθήσει και ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας. Έχουμε ένα πρώτο αριθμό τέτοιων project στην διαδικασία και σε όλη τη διάρκεια του χρόνου τα project αυτά θα εξυπηρετήσουν τον σκοπό της ευαισθητοποίησης των νέων σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Όταν είδαμε τα ανησυχητικά συμπεράσματα της μελέτης που σας ανέφερα, αποφασίσαμε να συντάξουμε ένα είδος βαθμολόγιο για να παρακολουθούμε ετησίως ή και αναεξάμεινο την εξέλιξη και να δούμε πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε πλησιότερο τους νέους και μέσα από ποιους διάβλους επικοινωνίας. Ορισμένοι από εμά γνωρίζουν καλύτερα τη χρήση των κοινωνικών μέσων. Περνούμε μέσα από τα κοινωνικά μέσα για να έλθουμε σε επαφή με τους νέους. Γιατί είναι και τα μέσα επικοινωνίας τα οποία ε, ε, απασχολούν πολύ τους νέους. Αλλά περνούμε μόνο θετικά μηνύματα γιατί γνωρίζουμε ότι οι νέοι αντιπαθούν τα αρνητικά μηνύματα. Ε, δηλαδή προβάλλουμε θετικά παραδείγματα όπου η πνευματική διοκτησία προσέφερε κάποια ωφέλεια σε έναν νέο δημιουργό ή σε κάποιον άλλο. Έχουμε λοιπόν αυτή την ιστοσελίδα που λέγεται Ideas Power, η δύναμη των ιδεών μπορεί να ενδιαφέρει αυτό του νέου. Έχουμε πολλές σχετικέ πρωτοβουλίες και μάλιστα σκεπτόμαστε και να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε ακόμα και νεότερους από το ηλικιακό φάσμα που αναφερθήκατε. τα πρόσωπα, τα, ε, ε, έχω εγώ λοιπόν ε, τα δικά μου τα παιδιά που έχουν και μεγάλη διαφορά μεταξύ τους έχουν ωστόσο πολύ μεγαλύτερη και ταχύτερη κατανόηση των θεμάτων αυτών από ότι εγώ. Για την κυρία Τρίπελ. Τι ακριβώς είπατε στην ερώτησή σας. Νομικές υπηρεσίες ποιότητος νομίζω είπατε. Αγαπητή κυρία Τρίπελ, υπάρχει, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι υπάρχουν κάποιες ε, νομικές υπηρεσίες που μπορούν να ανακόψουν αυτό το downloading. Για το 2013, αυτό το κομμάτι άφησα έξω, ε, εκτός της ομιλίας μου, το 2013 το ερευνητικό Ινστιτούτο Ήψους βρήκε ότι εκείνα τα χρόνια το παράνομο downloading κινηματογραφικών ταινιών και ε, τηλεοπτικών παραγωγών στην Νορβηγία μειώθηκε κατά το ίμιση. Και αλλού μειώθηκαν σημαντικά. Και το ύψους, το Ινστιτούτο λέει, επισημαίνει την δημιουργία άλλων εναλλακτικών επιλογών, όπως τα προγράμματα Netflix και Spotify για μουσική, το δεύτερο για ε, ταινίες το πρώτο. Είναι δηλαδή τα νόμιμα κανάλια. Αυτά ακόμα είναι εμβαλωματικά. Όπως είπατε και εσείς όμως, εκεί σημειώνονται σημαντικές αλλαγές και μάλιστα πολύ ταχείες. Αλλά βεβαίως όλες οι χώρες δεν είναι ισότιμες σε ό,τι αφορά το προσφερόμενο περιεχόμενο. Content δηλαδή. Αυτό μπορεί να φέρεται σε διαφορετικούς λόγους μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ισότητα στην πρόσβαση είναι σημαντικό θέμα όταν, όταν ε, ε, εξετάσουμε αυτό το βαθμολόγιο που έλεγα προηγουμένως και που μας δείχνει ότι 30% των νέων δηλώνουν ότι αυτό που τους οδηγεί στις παράνομες πηγές περιεχομένου είναι ότι αυτές είναι πιο εύκολο να τις βρουν και ταχύτερο το κατέβασμα. Και μάλιστα αυτούς, αυτά τα επιχειρήματα τα επικαλούνται συχνότερα γυναίκες από άνδρες. Αυτό δείχνει ότι είσαστε και πιο λογικές. Υπάρχει δηλαδή καθαρά μια διασύνδεση με την λογική. Για να απαντήσω στην ερώτησή δηλαδή, ναι, τα αποδεικτικά στοιχεία δεν είναι πλήρη, αλλά υπάρχει μια σαφή στάση. Αποτελεσματικό κόστος, πρόσβαση, ε, νομική, νόμιμες προσφορές ε, επηρεάζουν την πρόσβαση των νέων. Ε, δεν έχουμε τίποτα που να μας πείθει για το αντίθετο. Όσον αφορά τα υπόλοιπα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, κάνουμε ό,τι μπορούμε και αυτό συνδέεται με την αρχική μου παρουσίαση, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τις αρχές επιβολής του νόμου να καταπολεμήσουν την παραποίηση. Και όπως είπα, εμείς δεν είμαστε αρχή, ούτε πολιτικός οργανισμός, πολιτικό σώμα, αλλά αφιερώνουμε όλα τα μέσα που έχουμε ε, για να εξυπηρετήσουμε τις ε, πολιτικές αρχές και τις αρχές επιβολής του νόμου για να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Αυτά, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει ο κύριος Γραμματικάκης που ζήτησε τον λόγο, παρακαλώ. Γιώργης, μικρόφωνο. Okay. Οκ. Οκ. Ε, η ερώτησή μου έχει να κάνει με την ερώτηση της Προέδρου εσάς ε, κυρία Πρόεδρος γιατί νομίζω ότι απαντήθηκε με πολύ θα έλεγα μη ικανοποιητικό τρόπο. Ε, λέει ο μελετητής ότι κατά κάποιο τρόπο είναι λίγο ανεξάρτητη αλλά δεν είναι και πολύ ανεξάρτητη γιατί έχει και 10 ευρωβουλευτές μέσα εγώ δεν το ήξερα πρέπει να πω και ένα σεβαστό προϋπολογισμό μέσα στη δυσκολία που ζούμε όλοι ε, πρέπει να πω ότι η έκθεση του παρατηρητηρίου πάω σε άλλο θέμα τώρα, αλλά νομίζω εκεί θα ήθελα μια παραπάνω διασάφηση. Το ρόλο σας, τις σχέσεις σας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κλπ. Πάω σε ένα άλλο θέμα, γιατί ομολογώ ότι εντυπωσιάστηκα από τη μελέτη ως προς δύο-τρία στοιχεία και τη θεωρώ πολύ ενδιαφέρουσα. Το πρώτο είναι ότι από ό,τι θυμάμαι το 38% των νέων που χρησιμοποιούν παράνομη ιστοσελίδες όπως ταινίε το είπατε κι εσείς, 38% θεωρούν δεν κάνουν κάτι λάθος, εφόσον το υλικό προορίζεται για προσωπική χρήση. Δεν περνάει από το μυαλό τους δηλαδή καθόλου ότι μπορεί έτσι να θίγονται οι καλλιτέχνες και οι άνθρωποι που έχουν τη δημιουργική αυτή δραστηριότητα. Δεύτερο εντυπωσιακό νούμερο, ότι το 35% περίπου των νέων πιστεύει στους θελίδες που εμφανίζονται στα αποτελέσματα μιας μηχανής αναζήτησης είναι και νόμιμες. Αυτό ομολογώ μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση, δηλαδή είχα τους νέους ανθρώπους πιο ευφύς από εμά τους οριμότερους, δεν μπορεί πραγματικά να έχουν τέτοια παρεξήγηση. Και το ερώτημά μου είναι αυτό που επανέρχεται σε όλους τους συναδέλφους και το λένε πολύ καλύτερα από μένα. Τι μέτρα σκοπεύει να πάρει το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο με τις δικές του δυνάμεις για την παραβίαση αυτή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Είπα ότι δεν έχετε νόμιμες, νομικές έτσι δυνατότητες, αλλά το πρόβλημα παραμένει. Η δίκαιη αμοιβή των καλλιτεχνών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ε, Ευχαριστώ Γιώργο. Έχουν ενδιαφέρον αυτές οι ερωτήσεις, παρακαλώ απαντήστε. The observatory follows the model of governance of the agency. Πρέπει να δει κανείς τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η υπηρεσία αυτή. Ε, εμείς είμαστε αυτοχρηματοδοτούμενοι. Το παρατηρητήριο έχει λοιπόν, το UIPO έχει επίσης εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα και ε, εκπροσώπους των κρατών μελών εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκπροσώπους δικού σας. Αυτό είναι το πρότυπο διακυβέρνησης να το πω έτσι. I would not qualify whether the youngsters are stupid or not um, Τώρα για το αν είναι έξυπνοι ή όχι οι νέοι αυτό ε, δεν μπορώ να το πω εγώ αλλά πάντως τα αποτελέσματα που έχουμε μπροστά μας δεν δείχνουν μια καλή κατάσταση και αν το αφήσουμε έτσι όπως έχει το πράγμα τότε θα χειροτερεύσει η κατάσταση και αυτό σίγουρα όπως είπατε θα βλάψει τους καλλιτέχνες, τους δημιουργούς Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Εμείς δεν έχουμε εφαρμοστικές εξουσίες. Δεν είμαστε δύναμη καταστολής. Έχουμε όμως την δυνατότητα να φέρουμε στην επιφάνεια τις καταστάσεις αυτές. Κάναμε μια μελέτη στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να κατανοήσουμε πώς από τη μία η φαντασία και η δημιουργία και από την άλλη η προστασία της φαντασίας και της δημιουργίας μπορεί να διδαχθεί στα σχολεία χρησιμοποιώντας τις τις βέλτιστες πρακτικές από χώρες όπως η Νότια Κορέα και οι Ηνωμένε Πολιτείε και κάποιες σκανδιναβικές χώρες. Εμείς συνεργαζόμαστε με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την υπηρεσία της Επιτροπής την υπεύθυνη για την εκπαίδευση και δημιουργήσαμε δύο δίκτυα. Ένα δίκτυο για τους νέους και ένα δίκτυο για τους διδάσκοντες. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα είναι ενδιαφέροντα εκεί. Εμείς επίσης δημιουργούμε ένα σύνολο ε, νομικών ρυθμίσεων διαθεσίμων έτσι ώστε να γνωρίζουν ε, οι πολίτες που μπορεί να κατεβάσουν ε, εν πάση περιπτώσει νομίμως υλικό δεδομένα. Και είναι και κάτι το οποίο κάνουμε, ένα FAQ δηλαδή ε, επανειλημμένα ερωτήσεις γύρω από το θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας. Πολλές ερωτήσεις για ένα πράγμα βέβαια το οποίο είναι περίπλοκο ε, γιατί υπάρχουν 20 διαφορετικά καθεστώτα και είναι περίπλοκο το θέμα για μένα πόσο μάλλον για τους νέους των 12, των 14 και των 16 ετών βάση περιπτώσει προσπαθούμε με τα μέσα που έχουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Η ευθύνη όμως για τη λήψη μέτρων είναι περισσότερο στους δικούς σας όμως και όχι στους δικούς μου. Και σίγουρα έχουμε τις δυνάμεις που έχουμε πέραν αυτού σας ευχαριστώ. Κανένας δεν λέει ότι δεν πιστεύει ότι είσαστε νομοθετικό σώμα. Κανένας δεν λέει δεν πιστεύει ότι είσαστε αστυνομικό σώμα. Όμως η δική σας επαϊωσύνη, οι μελέτες, η δουλειά την οποία έχετε κάνει μέχρι τώρα στον τομέα της παραχάραξης και της παραποίησης και της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας δείχνει ότι πολλά μένει να γίνουν οι κατευθύνσεις σας βασίζονται σε τεκμήρια. Προσπαθείτε εσείς να κρατήσετε μια ισορροπία ανάμεσα σε ένα προφίλ προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας όχι μόνο σαν προστασία οικονομικών συμφερόντων, αλλά προστασία της δημιουργικότητας και να δημιουργήσουμε και νέα πρότυπα χρήσης του υλικού αυτού των δεδομένων αυτών έτσι ώστε να μην υπάρξει απομόνωση. Θα υπάρξουν ε, ίσως και περαιτέρω ε, ε, ερωτήσεις για διευκρινήσεις. Όταν έχετε περισσότερα τεκμήρια παρακαλώ να μας τα στείλετε. Το θέμα το κρατάμε ανοιχτό, δεν είναι η τελευταία φορά που σας συναντάμε και τίθεται αυτή τη στιγμή ένα ερώτημα ε, ε, είχα ζητήσει ποιος ε, θέλει το λόγο και καθυστερήσατε να απαντήσετε. Θα ήθελα λοιπόν μισό λεπτό να δώσω το λόγο στον κύριο Νεκόφ, ο οποίος ζήτησε με καθυστέρηση να πάρει το λόγο και αμέσως μετά θα ακούσουμε ένα σχόλιο της Επιτροπής και τη δική σας τελική απάντηση. Ευχαριστώ. Εκτιμώ πολύ το έργο σας. Ως νέος έχω μια ερώτηση. Πώς προτίθεστε να αντιστρέψετε την τάση στην χώρα μου, την Βουλγαρία, οι νέοι θεωρούν ότι το παράνομο downloading είναι πολύ ευκολότερο από το νόμιμο και γι' αυτό προσφέρουν σε αυτό. Οι νέοι που κατεβάζουν ταινίες με παράνομο τρόπο από ιστοσελίδες torrent δεν έχουν άλλωστε καμιά εγγύηση ότι αν πάνε στις νόμιμες θα φτάσουν τα χρήματα στους πραγματικούς δικαιούχους, δηλαδή τους καλλιτέχνες και δεν θα πάνε σε κάποιους οργανισμούς ή σε κάποιες οργανώσεις που διαβιώνουν στην σκιά. Για αυτούς το παράνομο κατέβασμα είναι πολύ ευκολότερο από το νόμιμο. Ευχαριστούμε. Να ακούσουμε και την Κομισιόν. Ε, συνοπτικά παρακαλώ. Και μετά να κλείσουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Ε, επί των όσων είπε ο Πρόεδρος της ΟΧΕΜ, οι πληροφορίες που παρέχει το παρατηρητήριο είναι πληροφορίες κλειδί για μας ε, για τη χάραξη πολιτικών σε αυτόν τον τομέα. Αυτή τη στιγμή η αναθεώρηση και η αξιολόγηση της οδηγίας για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής διαδιοκτησίας ε, βασίζονται σε αυτά. Οι ερευνές τους λοιπόν μας βοηθούν να πραγματοποιήσουμε αξιόπιστη εκτίμηση αντικτύπου για την αναθεώρηση αυτή. Επίσης, ναι, το παρατηρητήριο πράγματι δεν έχει νομοθετικές ε, εξουσίες, αλλά όταν κάνουμε μια προσπάθεια εναρμόνισης των δικτύων ε, και των αρχών των κρατών μελών από κάτω προς τα πάνω, επηρεάζει τα πράγματα σημαντικά. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, έχουν γίνει πολλές εκστρατείες ευαισθητοποίησης στο παρελθόν, μεταξύ κρατών μελών, με διάφορους τρόπους. Το κακό είναι ότι η αρνητική ενημέρωση δεν λειτουργεί, αλλά χρησιμοποιήθηκε εντατικά. Και θα δείτε ότι αναπτύσσονται τώρα στην ιστοσελίδα νέε εκστρατείε, πολύ ενδιαφέρουσε προ του νέου, αλλά δείχνοντα τα θετικά, τι θετικέ πτυχέ ε, των ε, δικαιωματών διονυτική ιδιοκτησία. Και κάτι τελευταίο, το είπε κάποιο μέλο, εγώ συμφωνώ όχι από προσωπική εμπειρία, ότι οι νόμιμε τοποθεσίε. Ε, μπορεί να είναι πιο περίπλοκες από τις παράνομες. Ο λόγος είναι απλός, διότι οι παράνομες τοποθεσίες βάζουν όλα τους τα χρήματα στο σχεδιασμό τους. Γι' αυτό είναι πιο απλές. Και εμείς ε, διαρκώς ε, το τονίζουμε, βασιζόμενοι στα δεδομένα που λαμβάνουμε από το παρατηρητήριο, ε, πρέπει να καταπολεμήσουμε τους, αυτούς που προσφέρουν τις παράνομες ιστοσελίδες και όχι τους χρήστες τους. Τα νούμερα, όπως ξέρετε, είναι εντυπωσιακά. Αν δούμε τα πόσα χρήματα κερδίζουν οι ιδιοκτήτες παράνομων ιστοσελίδων, ειδικότερα μέσω εσόδων από διαφημίσεις, και εμείς συνεργαζόμαστε και σε αυτό το τομέα με το παρατηρητήριο και με τα κράτη-μέλη για να δούμε πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τις βελτιστές πρακτικές και στους διαφημιστές ε, ώστε να βέβαια, ε, τους ε, αποθαρρύνουμε από το να διαφημίζονται σε τέτοιες τοποθεσίες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Πολύ ενδιαφέροντα τα σχόλιά σας. θα μπορούσε να γίνει κάποιο διαγωνισμό δημιουργικών νέων που θα μπορούσαν να επανασχεδιάσουν τι ιστοσελίδε έτσι ω θετική αντιμετώπιση έτσι να αποκτήσουμε και κάποιους δημιουργικούς νέους ε, μέσω της παραποίησης. Ε, μέχρι ένα σημείο φυσικά. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο για να κλείσετε τη συζήτηση. Ναι κυρίες και κύριοι, απλά για να απαντήσω μερικά στοιχεία. Οι νέοι που κατεβάζουν παράνομα, ναι, φοβούνται όμως τι μπορεί να τους συμβεί, υπάρχει επιβλαβές λογισμικό, ε, κλοπή ε, στοιχείων, ε, υπολογιστών, πιστοτικών καρτών όταν έχουν και φυσικά εμείς τώρα κάνουμε μια προσπάθεια να προσδιορίσουμε τα ποσοστά τέτοιων ιστοσελίδων όπου υπάρχει κίνδυνος προσβολής ενός προσωπικού υπολογιστή. Έχουμε και στοιχεία τα οποία μπορούμε να δώσουμε στους νέους και να τους πούμε ότι ο κόσμος αυτός δεν είναι τέλειος. Αντιθέτως ε, ε, ε χαρακτηρίζεται από πολλούς κινδύνους. Δεύτερον, η ΟΧΙΜ κάνει ό,τι μπορεί για την καταπολέμηση της παραποίησης. Έχουμε ένα μνημόνιο συνεννόηση με την Ευρωπόλ. Πρόκειται να υπογράψουμε ένα με τη Eurojust και θα χορηγήσουμε μισό εκατομμύριο ευρώ στην Ευρωπόλ για να δημιουργήσουμε ένα κέντρο συντονισμού για την καταπολέμηση των, της παραβίασης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο. Αυτό είναι ένα από τα μέτρα. Αυτά είναι κάποια από τα μέτρα που ακολουθούμε. Ευχαριστούμε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Μην διστάζετε να μας στέλνετε ό,τι θεωρείτε χρήσιμο, ειδικότερα για τον τομέα ε, της δημιουργίας ε, που μας απασχολεί και μας, και μας ενδιαφέρει ως Επιτροπή, ο οπτικοακουστικός τομέας, ε, γενικότερα βέβαια και στο θέμα της παιδείας το να βρούμε θετικές διαδικασίες για να βοηθήσουμε την όλη διαδικασία θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα ωφέλιμο. Τα στοιχεία που μας δώσετε προηγουμένως για μας είναι πολύτιμα. Αν δεν έχετε αντίρρηση λοιπόν ναι, βέβαια, μα στείλατε κάποιο υλικό. Αν συμφωνείτε, μπορούμε να το μοιράσουμε στου συναδέλφου. Αλλά α κρατήσουμε ανοιχτό το διαβλό επικοινωνία μεταξύ μα ε, και αν τα καταφέρουμε μια μέρα να έρθουμε και να σε επισκεφθούμε στο Αλικάντε. Ευχαριστώ πολύ. Bene, colleghi, qui continuiamo con i nostri lavori. Ας συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Έχουμε το σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης, την ανταλλαγή απόψεων με τον εισηγητή Ανδρέα Μπόξορ όσον αφορά την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τους νέους. Όπως γνωρίζετε, αυτή είναι η στρατηγική 10-18 που επαναξιολογείται κάθε τρία χρόνια. Αυτό είναι μια ευκαιρία ε, όχι απλά για να ανοίξουμε ένα διάβλο επικοινωνία με τη νέα γενιά όπως έπραξαν μέσω διαβουλεύσεων άμεσων και ο εισηγητής και ο συνεισηγητής αλλά όπως γνωρίζουμε εμείς έχουμε τεράστια ευθύνη ε, όσον αφορά τις πολιτικές των νέων. Ε, πρέπει να τις προσανατολίσουμε περισσότερο ώστε να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους, να φέρουν αποτελέσματα και να ανταποκρίνεται στις προτεραιότητες της Ευρώπης. Ε, όχι λοιπόν μόνο σε ε, πολύ συγκεκριμένους τομείς, αλλά γενικότερα. Όπως μας ζητούν οι νέοι, δίνω το λόγο στον συναδελφό Μπόξερ για την παρουσίαση αυτή. Και μετά θα δώσω στο λόγο στους Κιώδης και μετά σε όποιον τον ζητήσει. Παρακαλώ, Ανδρέα. Thank you very much, And I switch to Hungarian. Θα ομιλήσω την Ουγγρική. Μιλώ για το ανθρώπινο δυναμικό που είναι πολύ σημαντικό για την, ε, για την Ευρώπη και για το μέλλον της. Πρέπει να φροντίσουμε ώστε το δυναμικό αυτά τα 90 εκατομμύρια νέων στην Ευρώπη να μπορέσει να αποδώσει. Η οικονομική κρίση έχει πλήξει μεταξύ άλλων και ιδιαίτερα τους νέους. Η απόσταση που χωρίζει πλέον τους νέους από την κοινωνική ζωή μεγαλώνει. Αισθάνονται αποκλεισμένοι και πολλοί από αυτούς ριζοσπαστικοποιούνται. Αυτή είναι η κίνδυνη που κρύβει αυτή η εξέλιξη. Είναι σημαντικό, εν πάση περιπτώσει, να συνεχίσουμε αυτή την πολιτική υπέρ των νέων. Γνωρίζουμε ότι η πολιτική για τους νέους είναι υπόθεση αρμοδιότητας των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προσφέρει ένα πλαίσιο και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κονδύλια του λεγόμενου ανοιχτού συντονισμού, δηλαδή μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μπορούν να καθορίζονται στόχοι για την στρατηγική υπέρ των νέων και οι χώρες μέλη στη δική τους πλέον αρμοδιότητα μπορούν να αποφασίσουν ποια από τα εργαλεία αυτά θα χρησιμοποιήσουν και με ποιον τρόπο. Στην περίπτωση των κρατών μελών που οι δείκτες ε, είναι άσχημοι, όπου οι δείκτες είναι άσχημοι, πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέσα σε μεγαλύτερη κλίμακα. Είναι ξεκάθαρο ότι ποικίλουν τα προβλήματα από χώρα σε χώρα. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν ενιαία επίπεδα που να μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις χώρες. Πρέπει να εφαρμοστούν τα κατάλληλα μέσα ανα αναχώρα. Το στρατηγικό πλαίσιο της Ένωσης για την νεολαία φτάνει μέχρι το 2018 και αναφέρεται στην εκπαίδευση και κατάρτιση, το επιχειρήν, την υγεία, την συμμετοχή, τον εθελοντισμό, τους νέους στον κόσμο και την δημιουργικότητα και τον πολιτισμό. Αυτή είναι η επιμέρους τομείς. Η στρατηγική προβλέπει και δύο προτεραιότητες αφενός την διευκόλυνση της μετάβασης από το σχολείο στην επαγγελματική ζωή και αφετέρου την ένταξη στην κοινωνική ζωή στην περίπτωση νέων και ένα άλλο θέμα που διαπιστώνουμε πρόσφατα είναι βέβαια το γνωστό πρόβλημα της ρίζος που χρειάζεται να αντιμετωπιστεί. Όπως είπε η Πρόεδρος ήδη, η στρατηγική αυτή επανεξετάζεται ανά τριετία. Ο Γιώργος Παπανικολάου είναι αυτός ο οποίος ανέλαβε την τελευταία έκθεση, τη σύνταξη της εκθέσεως και εγώ αναλαμβάνω από ε, την σκητάλη από αυτόν. Τον Δεκέμβριο πέρσι τα θεσμικά όργανα συνέταξαν έκθεση για την υλοποίηση της στρατηγικής για την νεολαία και η έκθεσή μου βασίζεται σε αυτήν ακριβώς την μελέτη. Εξετάζω τα εθνικά μέτρα, εξετάζω τις πρωτοβουλίες στο επίπεδο της Ένωσης, έχουν διεξαχθεί και συναντήσεις με όλους τους ενδιαφερομένους κύκλους, και μέσα στα πλαίσια του Youth Forum με στόχο την συγκέντρωση πληροφοριών και δεδομένων για να βασίσω εκεί την έκθεσή μου. Υπάρχουν στατιστικές που δείχνουν τις τάσεις που σημειώνονται μεταξύ των νέων. Όσον αφορά την εκπαίδευση διαπιστώνονται θετικές τάσεις που παρόλα αυτά δεν μπορούν να κρύψουν τις πολύ μεγάλες διαφορές που υπάρχουν και μεταξύ των χωρών μελών σε ό,τι αφορά αυτούς που εγκαταλείπουν νωρίς το σχολείο εκεί σημειώνεται μια υπιστοδρόμηση στα νούμερα. Για, την, για τις ηλικίες 18-24 ετών ήταν της τάξης του 11,5% ο μέσος όρος. Σε ορισμένε χώρε όμω, όπω για παράδειγμα λε, το ποσοστό είναι υψηλότερο. Σημειώνω πάντω ότι οι σημερινέ νέε και νέοι είναι πολύ καλύτερα εκπαιδευμένοι από ότι οι παλαιότερε γενναίε. Ο δε αριθμό των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει ανέβει αισθητά. Για τις ηλικίε 30 έως 34 ετών το 1 τρίτο διαθέτουν πανεπιστημιακό πτυχίο. Παρ' όλα αυτά, το ποσοστό των ανέργων πάλι μέσα στις ομάδες αυτές και των πτυχών δηλαδή είναι εξαιρετικά υψηλό. Κάτι το οποίο οφείλεται στο γεγονός ότι τα επιστημονικά τους προσόντα δεν συμβαδίζουν με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Χρειάζεται λοιπόν να γίνει προσπάθεια να προσεγγίσουν οι δύο αυτές τάσεις. Υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι διαθέτουν υπερβάλλοντα προσόντα για την απασχόληση που βρίσκουν τελικά. Υπάρχει και μια ομάδα που χρειάζεται περαιτέρω κατάρτιση. πολλές νέες και νέοι δραστηριοποιούνται και στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Το 2014 82% των νέων συμμετέχουν σε κάποια πλατφόρμα online ή σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο. Μπορεί να πει κανείς δηλαδή ότι οι νέοι ζουν κατά κάποιο τρόπο σε ένα παράλληλο κόσμο. Δεν σημαίνει αυτό ότι δραστηριοποιούνται πολιτικά. Πολλοί από τους νέους δεν προσέρχονται καν στις εκλογές για να ψηφίσουν. Τα δεδομένα του έτους 2014 δείχνουν ότι το μισό περίπου των νέων ανήκουν σε κάποια οργάνωση, λέσχη, δίκτυο. Αυτό είναι βέβαια μια θετική τάση και πάντως πρέπει να την ενισχύσουμε. σε τρόπο ώστε και η συμμετοχή στις οργανώσεις αυτές να συμβάλλει και σε μια κοινωνική ένταξη. Είναι σημαντικό για τους νέους να μπορέσουν να εξασφαλίσουν μια ποιοτική θέση απασχόλησης, να τους επιτραπεί δηλαδή αργότερα να είναι οικονομικά αυτόνομοι. Όντω έχει μειωθεί κάπω η ανεργία σε πολλέ χώρε μέλη. Όμω η ανεργία των νέων εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό πρόβλημα. το υψηλότερο ποσοστό που είχε επιτευχθεί, που <laughs> εντό εισαγωγικών μπορεί να το πηγαίνει αυτό, ήταν τη τάξη του 23,9%. Διαπιστώνουμε πάντως ότι σε ορισμένες χώρες μέλη εξακολουθεί η ανεργία αυτή να είναι υψηλότερη. Όπως είπα ήδη, ανέρχονται σε 90 περίπου εκατομμύρια οι νέες και οι νέοι στην Ευρώπη. Από αυτούς ένα 9% περίπου είναι μακρόχρονα άνεργοι. Ένα 13% εντάσσονται περίπου στην ομάδα εκείνη οι οποίοι ούτε εργάζονται ούτε έχουν πτυχίο ή καν απολυτήριο γυμνασίου ηλικίου. Και εκτός αυτού υπάρχει και μεγάλος αριθμός νέων που απειλούνται από την φτώχεια και τον αριθμό αυτό τον υπολογίζω σε περίπου 27 εκατομμύρια. Αυτό οδηγεί σε μεγάλη περιθωριοποίηση όλο και περισσότερων νέων. Δυστυχώς. Δεν είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός των νέων που συμμετέχουν στην πολιτιστική ζωή. Θα έπρεπε λοιπόν καθήκον μας να είναι πρωτίστως να συμβάλλουμε ώστε οι νέοι να γίνουν ενεργά μέλη της κοινωνίας, να συμβάλλουν και στην οικονομική ζωή της κοινωνίας και ε, στην δημογραφική της εξέλιξη. Είναι καθήκον των χωρών μελών βεβαίω να δώσουν τη δυνατότητα στους νέους να δημιουργήσουν οικογένεια, να βρουν δουλειά με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων. Θεωρώ εξάλλου ότι για την αξιολόγηση της στρατηγικής για την νεολαία ε, διαγραφούν και πορείες προς το μέλλον. Χρειαζόμαστε δηλαδή προτάσεις για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να μειώσουμε την ανεργία των νέων, πώς θα βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των νέων, πώς θα βελτιώσουμε την ισότητα των ευκαιριών, πώς μπορούμε να φροντίσουμε ώστε να συμμετέχουν περισσότερο. Και βέβαια πώς μπορούμε να μειώσουμε την ριζοσπαστικοποίηση πολλών νέων. Ε, την ευθύνη φέρουν πρωτίστως οι χώρες μέλη. Ο συντονισμός είναι πολύ σημαντικός ωστόσο μεταξύ τους. Χρειάζονται συγκεκριμένα μέτρα οι χώρες μέλη, επαναλαμβάνω, είναι αυτές οι οποίες καλούνται να τα λάβουν. Η έκθεσή μου αυτά θέτει ως στόχους. Όσον αφορά την διάρθρωση του κειμένου μου, μέσα στο κείμενο θα φύγω τους διάφορους τομείς, θα ασχοληθώ με θέματα χρηματοδοτικών δυνατοτήτων για σχέδια υπέρ των νέων, θα μιλήσω και για το Erasmus ΣΥΝ, θα μιλήσω για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, για την πρωτοβουλία απασχόληση των νέων. Επίσης η έκθεσή μου θα αναφέρεται και στην ευθύνη των κρατών μελών και στα μέτρα που οφείλουν να λάβουν οι χώρες μέλη. Θα μιλώ για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας υπέρ των νέων, για την υλοποίηση της εγγύησης υπέρ των νέων που έχει θεσμοθετηθεί και πιστεύω πάντως ότι πρέπει να περιλάβω και κάτι για τα μέσα, τα εργαλεία εκείνα που θα μας επιτρέψουν να συμβάλλουμε στην τόνωση της απασχόλησης των νέων. για να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να βρουν δουλειά και να γίνουν ανεξάρτητοι. Γι' αυτό πρέπει, όπως είπα, να συγκλίνουν η εκπαίδευση και η κατάρτιση των νέων με τις ανάγκες της αγοράς. Αυτό μπορεί να γίνει με τη χορήγηση υποτροφιών μεταξύ άλλων. Εκτός, άλλων, εκτός των άλλων πρέπει να αποδώσουμε μεγάλη σημασία στην απασχόληση των νέων και στην απασχολησιμότητα των νέων. Όπως το κάνουν οι επιχειρήσεις. Εκεί πρέπει να βασιστούμε, στην προώθηση του επιχειρήν, με πρακτικές εξετάσεις, ε, με, συγγνώμη, με πρακτικές εξασκήσεις που μπορούμε να προσφέρουμε στους νέους. Αυτά θα τα λέω εγώ μέσα στο κείμενο της εκθέσεως μου. Επίσης ε, βέβαια θα ασχοληθώ και με την ενεργό συμμετοχή στην κοινωνική ζωή των νέων, όπως το είπα ήδη αυτό, διότι αυτή η συμμετοχή, όπως δείχνουν τα στατιστικά δεδομένα, είναι ανεπαρκής. Πιστεύω ότι οι νέες τεχνολογίες της επικοινωνίας πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να οθήσουμε τους νέους προς αυτή την κατεύθυνση. Άλλα σημαντικά πράγματα είναι βεβαίως η φροντίδα για την υγεία των νέων, ο και ένα τελευταίο να τονίσω κάτι ακόμη οι τοπικές και περιφερειακές οργανώσεις, ενώσεις αθλητικές ενώσεις κτλ χρειάζονται υποστήριξη Εδώ πρέπει να, να τονίσουμε κάποιες πτυχές. Τη συνεργασία ανάμεσα στην οικογένεια, το σχολείο και την εκκλησία, για παράδειγμα. Και να δημιουργηθεί ένας διαθρωμένος διάλογος με τις οργανώσεις αυτές. Το ίδιο πρέπει να συμπεριληφθούν στον διάλογο αυτών και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Thank you so much. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχουν πάρα πολλές πλευρές οι οποίες πρέπει να μας απασχολήσουν και να ενισχυθούν. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι βρισκόμαστε σε μια νέα φάση των σχέσεων με τους νέους. Αναφέρομαι στον διαφορετικό διάλογο έχουμε τη δυνατότητα συζήτησης, αντιπαράθεσης, κατά κάποιο τρόπο τους καθιστούμε εταίρους σε μια νέα φάση σχέσεων. Και έχει μεγάλη σημασία να δούμε ποια είναι τα κρίσιμα σημεία, τα δύσκολα σημεία αλλά και τα ισχυρά σημεία τα οποία μπορούν να μοιραστούν οι διαφορετικές γενιές μεταξύ τους, πώς μπορούν να, αξιοποιηθούν αυτές οι σχέσεις θα μου επιτρέψετε λοιπόν και εγώ να μπορέσω να συνεισφέρω σε μια σημαντική έκθεση. Λοιπόν θα δώσω το λόγο στους τρεις σκιώδεις, Νεκόφ, Τσαμπάσκι και μετά Μαραγάλ. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να έχω περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα χρόνο αυτή τη φορά ήμουν σκιώδης για την συγκεκριμένη έκθεση. Θα ήθελα λοιπόν και σαν σκιώδης αλλά και σαν νέος άνθρωπος να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Οι γνώμες των νέων στα πλαίσια μιας τέτοιας έκθεσης πρέπει να ληφθούν υπόψη. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι η έκθεση αυτή θα πρέπει να εξεταστεί και από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ της Νεότητας. Η ανάλυση την οποία παρουσίασε η συγκήτρια είναι κάτι το οποίο με βρίσκει σύμφωνο, αλλά μου επιτρέψετε όμως να κάνω και κάποιες επιπλέον προτάσεις. Πρώτον θα συμφωνήσω μαζί σας ότι δεν υπάρχει θα έλεγα συνεννόηση και συντονισμός ανάμεσα στην στρατηγική για τους νέους και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πολιτικές. Δεν υπάρχει κοινό πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στις διαφορετικές στρατηγικές και πολιτικές. Αυτό εκπλήσει γιατί η στρατηγική για τη νεότητα είναι πολύ σημαντική και έπρεπε να καλύπτεται ε, σωστά από τις υπόλοιπες. Οι οργανώσεις των νέων θεωρούν ότι οι απόψεις τους δεν λαμβάνονται υπόψη όταν καθορίζονται οι πολιτικές για τους νέους. Οι νέοι λοιπόν ενθαρρύνονται να λαμβάνουν πρωτοβουλίες, καταλήγουν σε γνωμοδοτήσεις οι οποίες όμως αγνοούνται. Συνέπως λοιπόν θα πρέπει να ζητήσουμε να υπάρξει περισσότερη επεξεργασία των θέσεων των νέων, να μας δίδουν τις απόψεις τους πάνω στις προτάσεις μας τις αρχικές, και να συνεχίζουμε το διάλογο μαζί τους. Υπάρχουν επίσης και κάποιες ανησυχίες εδώ συγκεκριμένες. Η ανεργία των νέων σαν παράδειγμα είναι πολύ πιο ισχυρή από ότι οι υπόλοιπες ε, μορφές ανεργίας. Επίσης ε, οι νέοι στις ε, νέες μεταναστευτικές ροές φύγονται φυσικά ιδιαίτερως από την κατάσταση αυτή. Η ενσωμάτωση των νέων δεν είναι κάτι το εύκολο βέβαια για αυτές τις κοινότητες και πάρα πολλοί νέοι καταδικάζονται να εργάζονται σε θέσεις απασχόλησης μη αντίστοιχες με τις ικανότητές τους. Για να βελτιώσουμε λοιπόν την απασχολησιμότητα των νέων θα πρέπει να ακολουθήσουμε νέες κατευθύνσεις, προτεραιότητες τα επόμενα τρία χρόνια. Πρώτον, θα πρέπει να επενδύσουμε σε οριζόντια απόκτηση γνώσεων όπως επιχειρηματικότητα, ξένες γλώσσες και κινητικότητα επίσης ήδη σε μία πρώτη φάση. Με τον τρόπο αυτό οι νέοι θα είναι πιο ικανοί και θα προσαρμόζονται καλύτερα σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Νομίζω ότι η απόκτηση των ικανοτήτων και οι μη ε, τυπικές ή παραδοσιακές μορφές εκπαίδευσης είναι πολύτιμες. Έχω εργαστεί στα πλαίσια της πρωτοβουλίας του δικτύου αλληλεγγύης Πήραμε λοιπόν την πρωτοβουλία να καταστήσουμε τις άτυπες μορφές εκπαίδευσης περισσότερο δημοφιλείς επιπλέον μέχρι και το 2018 ισχύουν ορισμένες συστάσεις σύμφωνα με τις οποίες τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν αυτά τα παράλληλα εκπαιδευτικά ε, συστήματα. Σε χώρες όπως η δική μου η Βουλγαρία τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Σε άλλες χώρες τα πράγματα είναι κάπως καλά. Πάντως έτσι θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε τις απαιτούμενες γνώσεις. Υπάρχει και το θέμα των μεταναστών που πολύ συχνά δεν έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις και ικανότητες. Εδώ νομίζω ότι οι άτυπες μορφές κατάρτισης θα βοηθήσουν, θα είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για την κοινωνική ενσωμάτωση των νέων που προέρχονται από μεταναστευτικές κοινωνίες. Αυτό θα πρέπει να είναι τμήμα της έκθεσης κυρίως της Επιτροπής Πολιτισμού. Η συνάδελφος αναφέρθηκε στα θέματα της επιχειρηματικότητας. Στον τομέα αυτό απαιτείται περισσότερη έμφαση ε, νομίζω ε, από ό,τι περιλαμβάνεται ήδη στην πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τσαμπάσκι έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ συνάδελφοι. τα προβλήματα που αναφέρεται με απασχολούν ιδιαίτερα και στην Ευρώπη οι ναι, νέοι αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Για πολλούς νέους ε, η μόνη λύση είναι η μετανάστευση. Σήμερα το πρωί μιλήσαμε για τη διαφύγη εγκεφάλων, brain drain. Θέλουμε να την αποφύγουμε. Πολλές στατιστικές έρευνες ε, καταδεικνύουν καθαρά την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω από 5 εκατομμύρια νέοι στην Ευρώπη κάτω των 25 δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι είναι προτεραιότητα η απασχόληση των νέων και ότι μελετά πολιτικέ για να διασφαλιστεί η απασχολησιμότητά του. Μία πολιτική είναι η εγγύηση για του νέου. Το Youth Guarantee, ένα μέσο με στόχο οι νέοι κάτω των 25 να λαμβάνουν κάποιες προσφορές για εκπαίδευση, για κατάρτιση, για δουλειά τέσσερις μήνες αφού ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Αυτό ακούγεται πολύ αισιόδοξο, αλλά η επιτυχία είναι αβέβαιη. Δεν πάει βέβαια να είναι ένα θετικό βήμα προς τα εμπρός. Τώρα, για να επιτύχουμε και να δώσουμε προοπτικές στους νέους, πρέπει να επιλέξουμε τις σωστές πολιτικές και να φροντίσουμε να εφαρμοστούν. Για να επιτύχει μια πολιτική πρέπει να υλοποιείται και να αναθεωρείται. Καλωσορίζουμε λοιπόν όλες τις εκθέσεις ε, υλοποίησης. Τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να ακούσουμε τους οργανισμούς νέων. Διότι αυτοί βρίσκονται κοντά στους νέους, γνωρίζουν τα όνειρα της φιλοδοξίας τους. Πρέπει να ακούσουμε τι τρόπους προτείνουν αυτοί για την επιλύση της κρίσης. Θα αναμένω με ανυπομονησία την έκθεση. Ε, το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Μαραγκάλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω όλη την παρέμβαση της εισηγήτριας. Νομίζω ότι αρκετά άκουσα πάντας. Άκουσα επίσης ε, τις πληροφορίες για τις τροπολογίες και τις συζητήσεις που θα έχουμε από εδώ και πέρα και θα, κάνουμε, θα κάνω μια γενική παρουσίαση. Υπάρχει μια έκφραση στα αγγλικά που εφαρμόζεται ίσως στην πολιτική των νέων που ακολουθείται στην Ευρώπη. Throwing money to problems, λέει ο μιλητής. Νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση όπως και να έχουν τα πράγματα για πάρα πολύ καιρό αυτό κάναμε. Νομίζω λοιπόν ότι και με τα, το Ταμείο για την Νεότητα και για την Πρωτοβουλία για τους Νέους ε, στην ουσία βλέπουμε αφού έχουμε δαπανίσει χρήματα ότι η απόσβεση, μάλλον η απόδοση των ταμείων αυτών είναι πάρα πολύ δύσκολο να φανεί είναι δύσκολο να δούμε θετικά αποτελέσματα παρά τα στοιχεία ε, τα οποία μας έδωσε και η συγγήτρια για τη σημερινή κατάσταση. Και αυτό ισχύει για πάρα πολλές ε, από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει εδώ να κάνουμε μία διευκρίνωση. Μιλάω για τα ευρωπαϊκά ταμεία, τα οποία προστίθενται θα έλεγα στο τι γίνεται σε κάθε χώρα. Αν θέλουμε να δούμε τι κάνουν και οι εθνικοί πόροι σε αυτή την περίπτωση, τότε πραγματικά θα μπορούσαμε να είχαμε την εικόνα της πραγματικής απόδοσης των επενδύσεων αυτών. Λοιπόν, Πρώτον, θα πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλύτερα αυτό το οποίο ισχύει και αυτό το οποίο εφαρμόζεται, να προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε κάπως καλύτερα, να ενισχύσουμε ταυτόχρονα τα προγράμματα τα οποία συνιστούν τις πολιτικές για την νεότητα. Δεύτερον, να πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάποιους κοινούς δείκτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όχι αυτούς οι οποίοι ε, θα έλεγα χρησιμοποιούνται ήδη, δηλαδή ποσοστό ανεργίας, πρόσβαση στην εκπαίδευση κτλ. Αλλά κάποια στοιχεία τα οποία θα επιτρέψουν να συνειδητοποιήσουμε μια καλύτερη εικόνα όχι ε, την κατάσταση ως έχει απλά, αλλά να προσπαθήσουμε να δούμε τι δυνατότητες έχει κάθε χώρα. Να καθορίσουμε επίσης κριτηρία μεγαλύτερης ευελιξίας και σωστής εφαρμογής της αρχής της επικουρικότητας. Γιατί κάθε χώρα και κάθε περιφέρεια θα μπορεί να εφαρμόζει με μεγαλύτερη ελευθερία, με μεγαλύτερη δυνατότητα, καλύτερες δυνατότητες τα μέτρα τα οποία θεωρεί πιο κατάλληλα, πιο προσαρμοσμένα για να καλυφθούν συγκεκριμένες καταστάσεις. Σαν παράδειγμα στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορέσαμε να δώσουμε ούτε ένα ευρώ επιπλέον στην European Youth Initiative. Εμείς έπρεπε να περιμένουμε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης την οποία θα πρέπει να διεξάγουν τα κράτη-μέλη σχετικά με την εφαρμογή των συγκεκριμένων ρυθμίσεων του ταμείου αυτού. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει καλύτερη ε, οργάνωση ως προς αυτό. Μεγαλύτερη λοιπόν ευελιξία, κοινοί δείκτες, πραγματική ολοκλήρωση ε, και συνδυασμός των δημοσιονομικών κοινοτικών μέσων με τους εθνικούς πόρους τότε θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε και τα προγράμματα συνοχής, σύγκλησης συγγνώμη, τα οποία οφείλει να εφαρμόσει κάθε χώρα μέλος έτσι ώστε να υπάρξουν θετικές αλλαγές σε τομείς όπως η απασχόληση, η παιδεία κτλ. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο η έκθεση αυτή θα μπορέσει να καταστεί χρήσιμη ως προς τις προτάσεις της. Έχω άλλους δύο που έχουν ζητήσει το λόγο. Σβεντρόβα και κάποιος άλλος συνάδελφος μετά θα ακούσουμε τον Επίτροπο, την Επιτροπή μάλλον, μετά τον εκπρόσωπο του Φόρουμ και μετά την εισηγήτρια. Μέσα σε 12 λεπτά όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομη διότι ο συνάδελφος περιέγραψε πολύ καλά την κατάσταση και τις ε, δυνατότητες και προτάσεις για το μέλλον. Δεν υπάρχει λοιπόν λόγος να επανέλθω στα ίδια, αλλά όταν αναφερόμαστε στην αποτελεσματικότητα των επενδυμένων ε, χρημάτων και κονδυλίων, έχουμε ήδη τις απαντήσεις. Ξέρουμε ότι το πρόγραμμα εγγύηση βοήθησε στη μείωση της ανεργίας. Ξέρουμε ότι το για παράδειγμα ότι το Εράσμους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Όσοι αποφύτησαν έχοντας κάνει εράσμους είχαν διπλάσια επιτυχία στην ευρύς θέση εργασίας. Γνωρίζουμε ότι οι απόφοιτοι που έκαναν εράσμους πηγαίνουν και ψηφίζουν. Το 80% πήγε ψηφίζει. Εμπλέκονται περισσότερο στην κοινωνία, στις ε, κοινότητες τους. Εάν τα προγράμματα λοιπόν ε, είναι καλά, τότε φυσικά είναι και αποτελεσματικά. Τώρα, εκτιμώ το ότι ε, αντιλαμβανόμαστε την ευθύνη που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τους Νέους και κάποιοι άλλοι οργανισμοί δραστηριοποιούνται ιδιαίτερα στον τομέα αυτό και αυτό αποτελεί επαρκή απόδειξη ότι η νέα γενιά κατανοεί, ε, βλέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως το δικό της χώρο ε, συμμετοχή, όπου μπορεί να δραστηριοποιηθεί. Κάτι πολύ σημαντικό για αυτού, ε, διότι όταν ε, εμείς ήμασταν νέοι τα πράγματα ήταν πολύ πιο περίπλοκα. Υποστηρίζουμε λοιπόν όσους προσπαθούν να δραστηριοποιηθούν, να φέρει αποτελέσματα και φυσικά θα πρέπει να παρακολουθούμε και το τι είναι αυτό που καθιστά αποτελεσματικά τα κονδύλια σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τρεις σύντομες συμπληρώσεις. Ήθελα να συμπληρώσω λίγο αυτά τα οποία είπε η κυρία Μπούτσκα. Αυτό που βρίσκω σημαντικό είναι ότι η νεολαία χωρίς την επικουρικότητα δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Δεν μπορούν να θεσπιστούν αυστηροί κανόνες για το μέλλον της νεολαίας. Μόνο συστάσεις μπορούμε να δώσουμε. Έχω και άλλα σχόλια. Πρώτο, οι τοπικές κοινότητες. Αφενός έχουμε την παγκοσμιοποίηση, τον έρασμο, πόσοι υποφελούνται από τον έρασμο, σε ποσοστό δηλαδή, είναι άλλη ιστορία. Όμως πρέπει να διαδικτυωθούν οι τοπικές κοινότητες. Αυτό είναι σημαντικό, διότι Δεν μπορούμε αλλιώς να εγγυηθούμε τις ρίζες των νέων. Εγώ έχω εργαστεί πολύ στον τομέα αυτό. Ειδικά με την κατεύθυνση που πρέπει να δούμε στους νέους. Όταν μιλούμε ως δάσκαλοι στους νέους έχει καλός. Όταν όμως οι νέοι φύγουν από το σχολείο και βεβαίω εκεί πέραν το μεγαλύτερο μέρο τη ζωή του ω ενήλικοι δεν έχουμε τόσους εμπειρογνώμονες για θέματα νέων. Πρέπει να στρέψουμε τα μάτια μας και σε αυτό το θέμα. Έχουμε ένα γερμανικό μοντέλο, έχουμε ένα σκανδιναβικό μοντέλο για τα πράγματα αυτά. Έχουμε βέβαια και τις αστυνομικές αρχές, αλλά δεν με απασχολούν τόσο αυτές. μένα με απασχολεί περισσότερο η πρόληψη και η συνεργασία μας βέβαια με τις αστυνομικές αρχές για την πρόληψη όμως πάντα. Και τρίτο, αλλά σημαντικό, να εξετάσουμε εάν μπορούν να σταθούν στα πόδια τους οι νέοι. Είναι διαφορετικό βεβαίως στα διάφορα κράτη-μέλη. Αλλά πώς θα μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους οι νέοι, πώς θα μπορέσουν να αναπτυχθούν να αναπτύξουν τις προσωπικότητές τους σε μια ανεξάρτητη ε, οικονομική και επαγγελματική ζωή. Αυτό είναι που πρέπει να περιληφθεί πρωτίστω στην έκθεση. Ευχαριστούμε τώρα. Δίνω το λόγο στην Επιτροπή. Παρουσίαση θα μας κάνει ο Τμήματάρχης ε, Πολιτικής για τους Νέους, Χαραλτ Χάριουτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εκ μέρους της Κομισιόν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους Κιώδης για την πολύ ακριβή απεικόνιση της κατάστασης των νέων και για την παρουσίαση των προτεραιοτήτων που θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Δεύτερον, επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω ότι η υλοποίηση μιας πολιτικής για τους νέους πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να υποστηρίζει και να συμπληρώνει τα όσα γίνονται σε εθνικό επίπεδο. Πού υπησέρχεται ο δικός μας ρόλος λοιπόν βοηθάμε στο συντονισμό ώστε να ενισχυθούν και να βελτιωθούν τα ατομικά ταλέντα των νέων. Και δεύτερον, για να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο οι νέοι με όλες τις προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν θα μπορούν να αναπτυχθούν. Για τον λόγο αυτό αναπτύξαμε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τους Νέους. Και με μεγάλη μας χαρά σας αναφέρουμε ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος. Να σας αναφέρω απλά που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις πληροφορίες. Έχουμε την έκθεση για τους νέους, αυτή καθεαυτή, και για όσους θέλουν να εμβαθύνουν. Έχουμε δύο έγγραφα εργασίας του προσωπικού της Επιτροπής για την κατάσταση των νέων, καθώς και για την υλοποίηση των πολιτικών για τους νέους ως ε, περαιτέρω αναγνώσματα και σύντομα θα υπάρχει διαθέσιμο online το Youth Monitor όπου θα έχουμε συγκεντρώσει δεδομένα ευρωπαϊκού επίπεδου ε, με, για τους 41 δείκτες για τους νέους και κατά κράτος μέλος. Του χρόνου θα έχουμε τα πρώτα κεφάλαια της ε, Wiki για τους νέους όπου θα λαμβάνετε επικαιροποιημένες πληροφορίες σε σχέση με την υλοποίηση των πολιτικών για τους νέους στις διάφορες χώρες. Ε, τα καλά νέα πιστεύω είναι ότι ε, στο πλαίσιο της στρατηγικής για τους νέους έχουμε καταφέρει πλέον σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη να έχουν ε, πολιτικές για τους νέους. Πρόσφατα 11 νέες χώρες ανέπτυξαν τέτοιες πολιτικές και σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο. Μάλιστα. Και αυτό θεωρώ είναι πολύ θετικό στοιχείο. Το δεύτερο νέο είναι ότι χρειάζεται είναι ότι έχουμε πλέον καταλήξει σε συμφωνία με το Συμβούλιο ότι στο πλαίσιο της στρατηγικής για τους νέους έχουμε τα τρία ετήσια ε, σχέδια εργασιών του Συμβουλίου όπου αναφέρονται οι προτεραιότητες με πρακτικά γεγονότα ε, για την Κομισιόν και σε εθνικό επίπεδο. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι τα εργαλεία που έχουμε αναπτύξει αρχίζουν να δείχνουν αποτελέσματα. Αλλά εξακολουθούν να χρειάζονται κάποιε μικρορυθμίσει. Να σα αναφέρω δύο στοιχεία τα οποία θεωρώ είναι σημαντικά. Πρώτον, και αυτό αναφέρθηκε από πολλούς ομιλητές, πρώτον λοιπόν η αναγνώριση των άτυπων και μη τυπικών δεξιοτήτων. Γεγονός που σημαίνει ότι αυτό που κάνουμε εμείς μέσα των δικών μας προγραμμάτων, αυτά που μαθαίνουν οι άνθρωποι ως εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, πρέπει να αναγνωρίζεται ώστε να μπορούν να βρουν εργασία. Έχουμε 500.000 ε, ε, διαβατήρια για τους νέους ε, τέτοιου είδους, αλλά οι επιχειρήσεις έχουν να κάνουν ακόμα πολλά για αυτά. Το άλλο που θα ήθελα να πω, κυρία Πρόεδρε, είναι το ζήτημα της συμμετοχής. Οι νέοι δεν συμμετέχουν πλέον τόσο πολύ στις παραδοσιακές μορφές δημοκρατίας, στις ψηφοφορίες, στις εκλογές. Αυτό είναι ένα κομμάτι του, μια πλευρά του νομίσματος. Η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι ότι οι νέοι ενδιαφέρονται για τα πολιτικά και θέλουν να συμμετέχουν, αλλά με τα εργαλεία που έχουμε αναπτύξει εμεί, τα εργαλεία που έχουμε αναπτύξει εμεί δεν του ενδιαφέρουν πλέον. Η πρόκληση λοιπόν είναι να του εκπαιδεύσουμε, να του καταρτήσουμε για εργαλεία τα οποία δεν του ενδιαφέρουν. Αντί γι' αυτό, θέλουμε να δούμε τι εργαλεία χρησιμοποιούν αυτοί οι ίδιοι και να τα προσαρμόσουμε στι δικέ του ανάγκε. Στο διαθρωμένο διάλογο λοιπόν θα αυξήσουμε και θα βελτιώσουμε την επικοινωνία και ε, σημειώνω αυτό που είπε ένα ομιλητή ότι αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να ενημερώνουμε καλύτερα τους νέους για το τι κάνουμε με τις ε, συστάσεις τους. Να τους δείξουμε ότι προσπαθούμε να βελτιώσουμε ε, τη δουλειά μας. Και κάτι τελευταίο. Ε, να αναφέρω την επικοινωνία, την πρωτοβουλία επικοινωνίας του Επιτρόπου μας ε, με νέου που κανονικά δεν συμμετέχουν σε αυτή τη δημοκρατική διαδικασία ώστε να τους δείξουμε ότι έχουν τη δυνατότητα να γίνει ακουστή η φωνή τους και να λάβουν σχολιασμό, να λάβουν ε, ενημέρωση. Αυτά κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που είπατε. Πραγματικά έχουμε τώρα μόνο πέντε λεπτά. Οπότε επειδή λαμβάνουμε στα σοβαρά τον διαρθρώμενο διάλογο, να ακούσουμε τον Τζον Βίλκεν που είναι εκπρόσωπος του European Youth Forum και μετά την εισηγήτρια έχουμε ελάχιστο χρόνο, αλλά ε, πρέπει οπωσδήποτε να ακούσουμε αυτούς τους ομιλητές. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χαιρόμαστε που τόσα μέλη της Επιτροπής ΚΑΛΤ έχουν δει την εκθεσή μας ε, και την έχουν διαβάσει. Αυτή συμπληρώνει το πολύ αναλυτικό έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι σημαντικό να διαμορφώνεται η πολιτική για τους νέους μαζί με τους νέους. Ε, σε, όλα τα στάδια χάραξη πολιτικής, από την αξιολόγηση μέχρι την υλοποίηση. Μόνο έτσι μπορεί κανείς να αξιοποιήσει τις επιτόπου εμπειρίες των νέων και των οργανισμών των νέων. Οπότε Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για τη συνεργασία με την Επιτροπή ΚΑΛΤ επί αυτή τη έκθεση, ώστε να δημιουργηθούν ακόμη περισσότερε συνέργειε μεταξύ διαφόρων στρατηγικών, ώστε η πολιτική για του νέου ε, να αποτελεί κομμάτι όλων των πολιτικών, να συντονίζονται καλύτερα οι εθνικέ πολιτικέ εν ώψη τη ε, υλοποίηση οροσύμων που θα επιτρέπουν ε, συγκρίσει σε εθνικό επίπεδο και με αυτόματη εμπλοκή των νέων και των οργανισμών για τους νέους σε όλα τα επίπεδα. Ε, κατά τη χάραξη πολιτική ξεκινώντας από το τοπικό επίπεδο το οποίο είναι και αυτό που βρίσκεται πλησιέστερα στους νέους ολόκληρης της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η συγγήτρια, οι ε, όπως βλέπετε, έχουν δείξει ότι έχουν διαβάσει προσεκτικά την έκθεσή σας. Υπάρχει αυτή η μέθοδος ε, το να προσπαθήσουμε να εργαστούμε λαμβάνοντας υπόψη το μέγιστο βαθμό της απαιτής σας. Δίνω το λόγο στην συναδέλφω στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ ε, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και όλες και όλους τους συναδέλφους μου καθώς και ιδιαίτερα βέβαια τους σκιοδισίτες για τις παρεμβάσεις τους, τις προτάσεις που μου υπέβαλαν και αναμένω βεβαίως με χαρά την συνεργασία. Εύχομαι και ελπίζω ότι θα είναι καλό το κείμενο που θα καταλήξουμε και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και το διάλογο με το Youth Forum. Eh, allora, il... Λοιπόν, η πρόταση η έκθεση θα παρουσιαστεί στις 18 και 19 Απριλίου και θα ακολουθήσουν οι κατάλληλες ημερομηνίες για τις τροπολογίες. Σας ευχαριστώ όλους, την εισηγήτρια, το Youth Forum και τους βουλευτές μας. Περιμένουμε λοιπόν φτάνει όπου να είναι ο Επίτροπος από τη μια στιγμή στην άλλη. Ε, μπορούμε να κάνουμε ένα πεντάλεπτο διάλειμμα. Ελπίζω όμως ε, ο αριθμός των συναδέλφων να αυξηθεί γιατί έχουμε συνάντηση με τον αρμόδιο επίτροπο. Πέντε λεπτά διάλειμμα.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

Dear colleague, Αγαπητοί συναδέλφοι, να ξεκινήσουμε. Καθίστε, παρακαλώ. Okay, uh, Ωραία, λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Είμαστε εντό των χρονικών ορίων. Ευχαριστούμε, κύριε Επίτροπε, για την επίσκεψή σας. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα αυτή η ανταλλαγή απόψε, αυτός ο διάλογος που συνεχίζεται και τώρα θα μιλήσω Ιταλικά. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που έχουμε εδώ τον Επίτροπο Ναύρατσετς ε, ως φιλοξενούμενο. Αυτή η τακτική ανταλλαγή απόψεων προβλέπεται στο πλαίσιο του διαρθρωμένου διαλόγου. Λίγο ησυχία παρακαλώ εκεί κάτω. Ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντικός ε, για εμάς Μεταξύ άλλων διότι η φετινή χρονιά θα επικεντρωθεί ελπίζω περισσότερο στα ζητήματα της εκπαίδευσης, της δημιουργικότητας των οπτικοακουστικών μέσων, της πολιτικής ε, για τους νέους. Το συζητήσαμε και προηγουμένως με την έκθεση της Επιτροπής μας. Όπως γνωρίζουμε στην ατζέντα και του Κοινοβουλίου και της Κομισιόν μας απασχολούν ε, οι προτάσεις που θα υπάρξουν και η δέσμευση του Επιτρόπου ε, για να δούμε και τι γίνεται μετά από τη διακήρυξη του Παρισιού. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Έχουμε αφιερώσει μια έκθεση σε αυτό για το διαπολιτισμικό διάλογο και την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης. Υπάρχει το θέμα της ατζέντα για τις νέες δεξιότητες στην Ευρώπη, New Skills Agenda for Europe, Θέλουμε οι πολιτικές εκπαίδευσης ε, να έχουν εκεί κεντρικό ρόλο, όχι μόνο η επαγγελματική κατάρτιση, διότι θεωρούμε ότι το μέλλον θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε με μια στιβαρή βάση πολιτιστική. Ξέρουμε ότι η Γενική Διεύθυνση ΕΜΠΛΕ και η Γενική Διεύθυνση Παιδεία συνεργάζονται στενά. Κάτι που μα χαροποιεί, διότι είναι σημαντικό να υπάρξει συντονισμό. Στι 24 Φεβρουαρίου οι Υπουργοί Παιδεία θα συζητήσουν το θέμα αυτό με παρόντε και του δύο επιτρόπου. Επίση, το σημαντικό θα είναι η Επιτροπή. Ε, σημαντικό θα είναι που θα ασχοληθεί η δική μας Επιτροπή και η Επιτροπή ΕΜΠΛΕ με παρουσία των δύο επιτρόπων αφού το ζητήσαμε εμείς. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να παρατηρηθεί κάποια έλλειψη ισορροπίας. Είναι σημαντικό επίσης και το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα δικαιώματα δημιουργού, για το copyright. Θα έχουμε την έκθεση φορητότητας που είναι η πρώτη πτυχή παρουσίαση παρουσίασε και εδώ θέλουμε να, να υπάρξει κοινή συνεργασία με την DG Connect Επίσης διαβάσαμε, διάβασα εγώ προσωπικά τις δηλώσεις του Επιτρόπου για αυτό το θέμα ότι το copyright δεν είναι πρόβλημα αλλά πόρος είναι κομμάτι της λύσης. Ελπίζουμε λοιπόν να ληφθεί αυτό υπόψη στα διάφορα προγράμματα της Κομισιόν και επίσης φυσικά ακούσαμε και την ανακοίνωση που θα ακούσουμε το Μάρτιο για τη νέα ευρωπαϊκή πολιτιστική διπλωματία. Από τους τρεις ε, επιτρόπους, την είπατε εκπρόσωπο κυρία Μογκερίνη, τον κύριο Ναύρατσιτ και τον Επιτρόπο Συνεργασίας και όλα αυτά μαζί με τις εργασίες που θα κάνουμε στο Κοινοβούλιο για την υλοποίηση των πολιτών προγραμμάτων. Όλα αυτά συνθέτουν ένα τεράστιο θεματολόγιο, σημαντικό θεματολόγιο για τη φετινή χρονιά μαζί με τα ζητήματα παιδείας ε, στο πλαίσιο του θεματολογίου για τη μετανάστευση. Οπότε μας ενδιαφέρει να μάθουμε από εσάς ε, για όλα αυτά τα συγκεκριμένα θέματα, τι έχετε να προτείνετε, ποια είναι η πρόταση της Κομισιόν, ποια η δέσμευση. Οπότε σας δίνω αμέσως το λόγο για 15 λεπτά όσα χρειαστείτε για να μας παρουσιάσετε το πρόγραμμα, να μας ενημερώσετε για τα τελευταία νέα και μετά θα δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους για ερωτήσεις και απαντήσεις. Ευχαριστούμε και πάλι που ήρθατε εδώ στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητά μέλη, κυρία Κώστα, απαριθμίσατε τα βασικά θέματα της εισαγωγικής μου ομιλίας. Γι' αυτό λοιπόν θα σταθώ λίγο πιο αναλυτικά σε κάθε ένα από αυτά Νομίζω ότι η συζήτηση της ημερήσιας διάταξης για τα επόμενα χρόνια είναι το πιο κρίσιμο χρονικά θέμα. Μαζί με την συνάδελφο Τάισεν επεξεργαζόμεθα την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απόκτηση επαγγελματικών ικανοτήτων έτσι ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες και τις αδυναμίες που υπάρχουν ε, βραχυπρόθεσμα και μέσο πρόθεσμα. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε επίσης ότι τα συστήματα κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσουν τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες και θα τους επιτρέψουν ε, να καλύψουν τις ανάγκες οι οποίες υπάρχουν. Στην παρούσα φάση τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης δυσλειτουργούν. Πάρα πολλοί ε, είναι αυτοί οι οποίοι δεν ολοκληρώνουν τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και δεν αποκτούν τις επιθυμητές ικανότητες. Αυτό παρεμποδίζει την δυνατότητα έντασής τους στις αγορές εργασίας. Η πρόκληση είναι να μην δώσουμε μόνο τις σωστές ικανότητες αλλά και τις σωστές στάσεις οι ε, ικανότητες όπως η δημιουργικότητα, η δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων, η κριτική σκέψη, όπως επίσης και ε, η δυνατότητα συνεργασίας είναι απαραίτητα. Ε, όσο ενωρίτερα κανείς νιώσει οικείος με αυτά, τόσο το καλύτερο. Πρέπει να ξεκινήσουμε στις τάξεις του δημοτικού η ανάπτυξη των ικανοτήτων πρέπει να συνοδεύει την φροντίδα των παιδιών από μικρή ηλικία. Πρέπει να συνοδεύει τα παιδιά στο σχολείο και να ολοκληρώνεται ε, μέσω της ε, κατάρτισης των ενηλίκων αργότερα. Εμείς λοιπόν δημιουργούμε μία ατζέντα η οποία βλέπει μακροπρόθεσμα και ξεπερνάει την απλή απασχολησιμότητα η Επίτροπος Τάισεν και εγώ συμφωνούμε πλήρως με αυτό και θα θέλαμε να προχωρήσουμε στον τομέα αυτό στη συνάντησή μας της 8ης Απριλίου. Ένα θα έλεγα η ικανότητα της επιχειρηματικότητας, της απόκτησης της επιχειρηματικότητας είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Θα βοηθήσει τους Ευρωπαίους να σταθούν μόνοι τους, να βελτιώσουν την αντοχή τους, να δώσουν νέα όθηση στο ομαδικό πνεύμα και την δημιουργικότητά τους. Η διδασκαλία της επιχειρηματικότητας θα είναι πολύ τιμή, όπως λέει και η έκθεση Σόιντρεβα οι σωστές επαγγελματικές ικανότητες θα βοηθήσουν τους πολίτες να βρούνε τις σωστές θέσεις απασχόλησης κατά του κοινωνικού αποκλεισμού. Χρειάζονται περισσότερα όμως έτσι ώστε να έρθουμε κοντά στους νέους και να βοηθήσουμε τις πιο εύθραυτες κατηγορίες να πέσουν στα περιθώρια της κοινωνίας ε, στην ε, ριζοσπαστική και βίαιη αντιμετώπιση των προβλημάτων. Εδώ και ένα χρόνο εγώ και οι Υπουργοί Παιδείας όλων των χωρών μελών αποφασίσαμε μέσω της εκπαίδευσης να προωθήσουμε τις αξίες αυτές. Πολύ σύντομα θα κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις έτσι ώστε αυτή η πολιτικά ανηλυμένη υποχρέωση να γίνει πραγματικότητα σε κοινοτικό, εθνικό και περιφερειακό τοπικό επίπεδο. Τώρα κάποιες από τις πρωτοβουλίες να σας παρουσιάσω. Πρώτον, θα ήθελα να εντατικοποιήσουμε τις ανταλλαγές ανάμεσα στα κράτη-μέλη των βέλτιστων εμπειριών. Ας πούμε το πρόβλημα της ριζοσπαστικοποίησης και της βίας στους νέους είναι ένα πρόβλημα συλλογικό και γι' αυτό ακριβώς οι πρωτοβουλίες που έχουν αποδώσει σε ορισμένες χώρες μπορεί να είναι χρήσιμες και στις υπόλοιπες. Δεύτερον, απαιτείται να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο με τα κοινωνικά ταμεία και τα κοινοτικά προγράμματα. Το Erasmus Plus παίζει καθοριστικό ρόλο. Έχω διαβεβαιώσει ήδη ότι τα επόμενα χρόνια 400 εκατομμύρια ευρώ θα είναι διαθέσιμα για προγράμματα προώθησης του σεβασμού της ιδιότητας του πολίτη και της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού. Στο τέλος του μήνα θα διατεθούν, θα ανακοινωθεί η διάθεση 13 ήδη εκατομμυρίων γι' αυτό. Η υποστήριξη των προγραμμάτων αυτών θα δοθεί στις πόλεις που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του κοινωνικού αποκλεισμού. Κάποιες πόλεις το χρειάζονται περισσότερο από ό,τι άλλες. Τρίτον, απαιτείται να επιταχύνουμε την υποστήριξή μας προς τους καθηγητές και διδασκάλους. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα απαιτούμενα μέσα με καλύτερο τρόπο. Σαν παράδειγμα το e-learning και οι online πλατφόρμες που συνδέουν 200.000 διδάσκοντες στην Ευρώπη πρέπει να διευρυθούν και προς τις γειτονικές χώρες που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα θέματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί επίσης να βοηθήσει και τις ιονή ανταλλαγές και επαφές μέσω του ηλεκτρονικού εράσμους. Θα ξεκινήσουμε φέτος με τη διασύνδεση 10.000 φοιτητών ε, στον τομέα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Θα υπάρξει επίσης ε, ε, ένα ειδικό βραβείο για αθλητικές ομάδες οι οποίες βοηθούν στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Πιστεύουμε ότι κάποια μοντέλα πρότυπα για την κοινωνία όπως αθλητές, καλλιτέχνες κτλ. μπορούν να πηγαίνουν στα σχολεία και να συμμερίζονται τις εμπειρίες τους με αυτούς με τους νέους. Επίσης πρέπει να ενισχύσουμε αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με τους νέους, τους κοινωνικούς λειτουργούς, διαμεσολαβητές κτλ. Παίζουν ένα τεράστιο ρόλο. Πρέπει να τους βοηθήσουμε να έχουν τις ικανότητες τις κατάλληλες για την αντιμετώπιση της ε, ριζοσπαστικοποίησης περαιτέρω θα ενισχύσουμε επίσης και την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία και θα την ανοίξουμε ε, σε ακόμα περισσότερους νέους που δεν έχουν πολλές δυνατότητες και ευκαιρίες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε ένα ψήφισμα πρόσφατα για τον πολιτισμικό διάλογο ε, και την προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και κυρίως την κυρία Julie Ward για μια πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια. Να στραφώ τώρα ε, στους μετανάστες και πρόσφυγες. Πρόσφατα έφτασαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ η εκπαίδευση έχει να παίξει σημαντικό ρόλο. Θα βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους να δουν τη θέση τους στις κοινωνίες μας προετοιμάζουμε μια σειρά πρωτοβουλειών για την υποστήριξη των μεταναστών και των προσφύγων και θα την την άνοιξη. Στο κέντρο θα είναι η εκπαίδευση. Πολλές χώρες μέλη ήδη έχουν ε, δημιουργήσει τα νομικά πλαίσια για την παροχή εκπαίδευσης στα παιδιά αυτά. Στην Ολλανδία ξεκίνησε, ή μάλλον η Ολλανδική Προεδρία ξεκινά μια πρωτοβουλία για την ανταλλαγή πρακτικών ανάμεσα στις διάφορες χώρες. Συνεργαζόμαστε επίσης ε, και με τα κέντρα αμοιβαίας αναγνώρισης τίτλων έτσι ώστε να δούμε τι εμπειρίες υπάρχουν για τη βοήθεια προς τους πρόσφυγες να συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους, να παίρνουν τα πτυχία τους και να αποκτούν επαγγελματικές ικανότητες το ταχύτερο δυνατόν. Μέσω του Erasmus Plus επίσης θα προσφέρουμε και μαθήματα online και θα δώσουμε τη δυνατότητα σε σε μετανάστες ε, επιστήμονες και πρόσφυγες επιστήμονες να συμμετέχουν σε προγράμματα όπως Μαρή Κιουρί και άλλα. Η προώθηση της αμοιβαίας διαπολιτισμικής κατανόησης είναι κάτι το βασικό. Πρέπει να ενισχύσουμε όμως τον διάλογο και με τους εταίρους μας στον υπόλοιπο κόσμο. Η πολιτιστική διπλωματία έχει να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Όταν μιλάω για τέτοιου είδους διπλωματία, μιλάω για αμοιβαία ε, ε, προσπάθεια εκπαίδευσης. Ε, έχουμε ήδη κάποιες εμπειρίες στον τομέα αυτό χάρη στη δική συστήριξη και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω δράσης στις εξωτερικές μας σχέσεις. Συνειδητοποίησαμε ότι πολλοί στον κόσμο ενδιαφέρονται ιδιαίτερα να εμπλακούν σε πολιτιστικό διάλογο με την Ευρώπη. Απαιτείται όμως μια πιο στρατηγική αντιμετώπιση του θέματος. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται για μια νέα στρατηγική στον τομέα των διεθνών σχέσεων μαζί με την ύπατη εκπρόσωπο κυρία Μογκερίνη θα δημιουργηθεί ε, θα έλεγα μια μορφή διπλωματίας πολιτιστικής η οποία θα δείχνει την εικόνα της Ευρώπης στον κόσμο, θα διευκολύνει τον διαπολιτισμικό διάλογο και θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την επικοινωνία μας βασισμένη στην εμπιστοσύνη. Οι πολιτιστικές ανταλλαγές θα πρέπει να είναι στο κέντρο φυσικά των προσπάθειών μας. Είναι αλήθεια ότι αυτές οι άμεσες επαφές ανάμεσα στους λαούς ε, βασίζονται σε αρχές και θεμελιώδεις αξίες. Θα συνεργαστούμε λοιπόν με κυβερνήσεις ε, και με πολιτιστικές οργανώσεις. Η στρατηγική μας δεν θα προσθέσει ένα επιπλέον στρώμα γραφειοκρατίας. Αντίθετα, θα μπορέσουμε να συμπληρώσουμε τις δραστηριότητες των κρατών μελών και να συνδυάσουμε τις δυνάμεις μας. Αρκετές πρωτοβουλίες έχουν ήδη ξεκινήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σαν παράδειγμα το πιλωτικό πρόγραμμα για τη στήριξη των δικτύων των νέων δημιουργικών εργοδοτών της Ένωσης με τρίτες χώρες. Εμείς κάνουμε προσπάθειες έτσι ώστε και το θέμα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς να αντιμετωπιστεί λόγω ακριβώς των λαιλασιών σε χώρες όπως η Συρία. Μαζί με τον συνάδελφο Μοσκοβισή Προσπαθούμε να βρούμε νομοθετικά μέτρα για την εισαγωγή των πολιτιστικών αγαθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, προσπαθούμε να βρούμε τον καλύτερο τρόπο χρήσης του αθλητισμού στην πολιτιστική διπλωματία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε μια ομάδα υψηλού επίπεδου για την λεγόμενη αθλητική διπλωματία ε, συγκεκριμένες προτάσεις τους καλοκαιρινούς μήνες. Ξέρετε ότι αυτά που μαθαίνουμε από τον αθλητισμό δεν είναι θετικά. Πάρα πολλά σκάνδαλα που έχουν θέσει σε κίνδυνο το αθλητικό ιδεώδες, προβλήματα με τα ναρκωτικά, με τις ουσίες, προβλήματα διαφορά στη FIFA κτλ. Εμείς έχουμε υιοθετήσει ένα ψήφισμα και εσείς σαν κοινοβούλιο μάλλον Επί τη βάση λοιπόν και της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρηστή διακυβέρνηση από τα διεθνή αθλητικά σώματα μικρά και μεγάλα να αναλάβουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις και ευθύνες και να μπορέσουμε έτσι να δούμε το τι πραγματικά γίνεται. Ένας άλλος τομέας στον οποίο θα κάνουμε προτάσεις είναι η πνευματική ιδιοκτησία με την προσπάθειά μας στον τομέα της ψηφιακή δημιουργικότητας νομίζω ότι θα απελευθερώσουμε τις ευρωπαϊκές ικανότητες. Πέρυσι ορίσαμε σωστά τους στόχους μας. Φέτος περνάμε σε δράση με νομοθετικές πρωτοβουλίες για ε, τις διάδοσης ε, του προστατευμένου από, από πνευματική ιδιοκτησία περιεχομένου. Έτσι θα μπορέσουμε και τη διάδοση του πνευματικού περιεχομένου να ενισχύσουμε και να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε τα μοντέλα προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας που βασίζονται στις, ε, στις αδειοδοτήσεις σε περιφερειακό επίπεδο. Νομίζω λοιπόν ότι οι προτάσεις αυτές έχουν σχέση και με, με την φορητότητα του περιεχομένου. Ταυτόχρονα θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η δημιουργία ε, θα πρέπει να προστατευτεί με δίκαιο τρόπο. Δηλαδή με την εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού για όλους και από αυτούς που υποφελούνται από το προστασία του copyright και βεβαίως προστασία των κατόχων του copyright. Δεν θα είναι εύκολη η επιτευχή του στόχου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει ακόμη διάφορες επιλογές. Αλλά σας λέω σαφώς ότι θα προσεγγίσουμε το θέμα με ισορροπημένο τρόπο, όπως εξηγήσαμε στην ανακοίνωσή μας για την οργάνωση του copyright πέρσι. Γι' αυτό και μου αρέσει το ψήφισμα προς την κατεύθυνση ενός ε, νόμου για την ψηφιακή αγορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πέρσι, που έχει τους ίδιους στόχους. Θα συνεργαστώ με τους συναδέλφους μου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και με εσά Ευρωβουλευτές για να επιτύχουμε τον κοινό αυτό στόχο. Θα ολοκληρώσω τώρα με λίγα λόγια σχετικά με την εφαρμογή των πιο σημαντικών προγραμμάτων μας. Erasmus, SIN και Creative Europe. Πολύ σημαντικά αυτά και στα πλαίσια της ε, ενδιάμεσης αναθεώρησης του ε, ε, δημοσιονομικού πλαισίου. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Χάρη και στις δικές σας προσπάθειες έχουμε δύο ισχυρά, καλά, γερά χρηματοδοτημένα προγράμματα που προχωρεί η εφαρμογή τους. Στον πρώτο του χρόνο ο Έρασμο ΣΥΝ στήριξε χρηματοδοτικά πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους και χρηματοδότησε 18.000 project. Το πρόγραμμα είναι και πιο ανοιχτό. Πάνω από 30% των 650.000 mobility funds για νέους πήγαν σε νέους που είχαν περιορισμένες ευκαιρίες. Τα νούμερα που μας έρχονται τώρα είναι πια για το 2015 και δείχνουν παρόμοια επιτυχία. Όπως είπα και πριν, φέτος θα δώσουμε προτεραιότητα σε project που προωθούν θεμελιώδεις αρχές, την κοινωνική διάσταση, την ενεργό συμμετοχή, και μια χείρα βοηθεία προ μετανάστε και πρόσφυγε. Έχουν υπάρξει και ορισμένα τεχνικά θέματα, αλλά συνεργαζόμαστε στενά με τι χώρε μέλη, ώστε το πρόγραμμα αυτό να γίνει πιο εύχριστο και πιο σταθερό. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε βελτιώσει του επόμενου μήνε. Το πρόγραμμα τώρα της Δημιουργικής Ευρώπης έχει φτάσει στην ταχύτητα κρουαζιέρας όπως λέμε. Το 2016 θα ξεκινήσουμε τον μηχανισμό χρηματοδοτικής εγγύσεω που θα προσφέρει σε επιχειρήσεις όλη την Ευρώπη ακόμα περισσότερες ευκαιρίες δίνοντας πρόσβαση σε τραπεζικά δάνεια εκτός από τι χορηγήσει του ίδιου του προγράμματος. Από την αρχή του φετινού χρόνου χρησιμοποιούμε την Creative Europe και για την στήριξη πολιτιστικών προγραμμάτων για την ένταξη των προσφύγων. Αγαπητά μέλη, σας διαβεβαιώ ότι ε, βασίζομαι σε εσά στην υποστήριξή σας για όλα αυτά, για την κοινωνική συμπερίληψη, ιδίως των νέων, που αυτή είναι η top προτεραιότητά μου και είμαι πεπισμένος ότι μαζί χέρι με χέρι μπορούμε να τα επιτύχουμε. Να δείξουμε στον κόσμο δηλαδή ότι επενδύουμε στους ανθρώπους. Αυτό θα είναι καθοριστική σημασία παράγοντας για την επίτευξη του, ε, για την επιτυχία μάλλον στο μέλλον είμαι βέβαιος ότι θα μας συνδράμετε. Την προηγούμενη εβδομάδα άρχισε η νέα φάση αυτού του νέου αφηγήματο για την Ευρώπη. Ενό project που ξεκίνησε εδώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα διεξαγάγουμε πολλέ συζητήσει ακόμη του επόμενου μήνε με του νέου και τι νέε. Και σα προσκαλώ να συμμετάσχετε. Πολύ ευχαρίστω τώρα θα ακούσω τι απόψει, σχόλια και ερωτήσει σα. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Πιστεύω ότι όλοι όσοι βρίσκονται εδώ εκτίμησαν το γεγονός ότι αυτό το βαρύ πρόγραμμα, το θεματολόγιο περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες προτάσεις. Βρισκόμαστε ενώπιν ενός προγράμματος δραστηριοτήτων δικό σας που μοιράζεται με άλλους επιτρόπους που ανταποκρίνεται στους στρατηγικούς στόχους η προσέγγιση μέσω της εκπαίδευσης και της δημιουργικότητας και της νέας γενιάς στην Ευρώπη. Θα πω εγώ τα δικά μου σχόλια αργότερα, να δώσω πρώτα το λόγο στους συναδέλφους που τον ζήτησαν. Ξεκινώ από τους συντονιστές, ε, η κυρία Φεραίεν πρώτα απ' όλα και μετά Καμερέβερτ. Πρώτα πρώτα σας ευχαριστώ. Πρώτα πρώτα για τον χρόνο που διαθέτεται στην Επιτροπή Πολιτισμού. Είναι σημαντικός αυτός ο διάλογος και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το τι πράττει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θεωρεί ότι μπαίνουν τα κέντρα βάρους. Ήταν πραγματικά ένα μεγάλο μπουκέτο θεμάτων αυτό που αναπτύξατε. Θα ήθελα παρόλα αυτά να τονίσω κάπως περισσότερο ένα θέμα το οποίο θίξατε ακροθυγώς στο τέλος, δηλαδή τα μοντέλα χρηματοδότησης στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα. Τα τελευταία χρόνια και σε άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές έχουμε μιλήσει και για το πρόγραμμα Horizon, για το FC και για όλα τα χρηματοδοτικά μοντέλα τα οποία υποτίθεται ότι θα εξυπηρετήσουν στην βελτίωση της χρηματοδότησης στην Ευρώπη και του δημιουργικού τομέα και εκεί μπαίνουν και όλες αυτές οι creative and cultural industries που είναι μία από τις αγορές που προσφέρουν σημαντικό δυναμικό ανάπτυξης. Εκεί συνεργάζεστε με την Μοέραση, με την Βιγέν Κόσκα που αναπτύσσουν επίσης στρατηγική στην χρηματοδότηση προγραμμάτων και περισσότερη χρηματοδότηση από όλα τα προγράμματα που χρηματοδοτούμε εμείς. Είναι βεβαίω τελείω διαφορετικά τα κονδύλια που μπορούν να διαθέτουν εκεί. Μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των διαφόρων δηλαδή επιτρόπων αναπτύσσεται τις αντίστοιχες στρατηγικές ώστε να προχωρήσετε εναρμονισμένα στην εξασφάλιση χρηματοδότηση για τον τομέα αυτό. Τώρα για το έρασμο συν. Τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία, καιρό μάλλον, έχουν διεξαχθεί διάφορες ε, ακροάσεις για το Ερασμοσύν που ε, τόνισαν τα όχι μόνο θετικά σημεία, υπάρχουν και αρνητικά. Υπάρχουν προγράμματα τα οποία δεν έχουν καμία ευκαιρία να ληφθούν υπόψη, ιδίω ε, για την ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση. Χρηματοδοτήσεις επίσης για τα σχολεία. Εκεί χρειάζεται πολύ περισσότερο συντονισμός. Αυτό βρίσκει σύμφωνη την Κομισιόν ή εν ώψη και των εξελίξεων που σημειώνονται στις κοινωνίες μας και της τάσεως προς ρίζος παστικοποίηση μήπως θα έπρεπε να προωθήσουμε πολύ περισσότερο αυτή την εργασία βάσης αντί να επισημαίνουμε τόσο πολύ αυτά τα εμβληματικά έργα όπως είπατε και εσείς και που καμιά φορά αυτό βλέπουμε κυρίως σε πολλές περιφέρειες της Ευρώπης. Για μένα ήταν πολύ θετικό το ότι θίξατε και το θέμα της μετανάστευσης και πώς είναι δυνατό μέσα από την εκπαίδευση, μέσα από την κατάρτιση, μέσα από την προσφορά γλωσσικών μαθημάτων να δώσουμε ένα χέρι βοήθεια στους ανθρώπους αυτούς που προσέρχονται στις ευρωπαϊκές κοινωνίες ως πρόσφυγες ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν καλύτερα ποιες είναι οι δυνατότητες, ποια είναι τα μέσα που μπορούν να δοθούν εδώ στην δουλειά βάσης που κάνουν οι κοινότητες, τοπικές κοινότητες για να μπορέσει να προχωρήσει αυτή η εργασία ένταξης των προσφύγων. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κάμερ Εβερτ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πραγματικά πολύ και εσάς κύριε Επίτροπε για την τοποθέτησή σας, για τις προτεραιότητες που εξηγήσατε Αρχίζω με την πολιτιστική κληρονομία με την οποία και εσείς ασχοληθήκατε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδίως εμείς ως Επιτροπή Πολιτισμού έχουμε στρατευθεί ώστε το 2018 να κηρυχθεί έτος πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη. Είναι περιορισμένος, ας το πω έτσι, ο ενθουσιασμός κυρίως στην ηγεσία της Κομισιόν διότι θεωρούν ότι αυτά δεν έχουν μεγάλη σχέση με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα μια τοποθέτηση δική σας. Γνωρίζουμε ότι τα κράτη-μέλη έχουν προχωρήσει σημαντικά τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υπόθεση αυτή και νομίζω ότι χρειάζεται πράγματι εδώ μια ταχεία λήψη αποφάσεως. Θα ήθελα να πω κάτι επίσης για την επανεξέταση του έρασμος ΣΥΝ. Η κυρία Βερχάιν είπε ήδη ότι ο έρασμος ΣΥΝ εξακολουθεί να είναι ιστορία επιτυχίας, χωρίς καμία αμφιβολία. Ωστόσο, σημειώνεται με ένας αριθμός προβλημάτων που δεν θα τα χαρακτήριζα ως μονάχα διοικητικά, διοικητικού χαρακτήρα. Θα έλεγα μάλιστα ότι εδώ υποσκάπτεται η εκδηλωμένη βούληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για να μην πω ίσως υποσκάπτεται εν πάση περιπτώσει ερμηνεύεται με διαφορετικό τρόπο ας το πω έτσι εμείς ζητούμε τα ονόματα των προγραμμάτων να παραμείνουν αναγνωρίσιμα. Είναι δηλαδή κατά κάποιο τρόπο σήματα κατατεθέντα τα οποία δεν επιτρέπεται να εξαφανιστούν. Διαπιστώνουμε όμως στις συζητήσεις με τους εθνικούς οργανισμούς που καλούνται να εφαρμόσουν τα προγράμματα ότι εξαφανίζονται σιγά σιγά τα ονόματα των προγραμμάτων αυτών και αντιμετωπίζουμε ξανά και ξανά κάποιους που λένε ότι το πρόγραμμα Κομένιους δεν υπάρχει πια. Κάτι το οποίο δεν ισχύει. Εμείς θέλαμε τα πράγματα αυτά να απλοποιηθούν. Ακούμε ωστόσο ότι οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων είναι ακόμα πιο δύσκολες. Καθόλου δεν ήταν αυτή η επιθυμία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτή η διαδικασία review που αρχίζει τώρα θέλουμε να εγγύψει ακριβώς σε αυτά τα προβλήματα και να εξεταστεί κατά πόσον αυτά τα οποία έχουμε όντως δηλώσει ως πρόθεσή μας στο παρελθόν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα όπως αυτή διαμορφώνεται στο πεδίο σήμερα. Έχουμε μιλήσει και για την ενδεχόμενη χρηματοδότηση προγραμμάτων γλωσσικών μαθημάτων. Βεβαίως, η ενσωμάτωση των προσφύγων στις κοινωνίες μας θα κοστίσει χρήματα. Είναι σαφές. Το ερώτημα είναι από πού θα πάρουμε τα λεφτά αυτά. Η μεγάλη δική μου ανησυχία είναι ότι τα λεφτά θα πάνε να τα βρουν εκεί όπου ούτω ή άλλω είναι περιορισμένα. Όταν ακούω δηλαδή για γλωσσικά μαθήματα από το έρασμο ΣΥΝ, αμέσως αναρωτιέμαι και από πού θα λείψουν τα λεφτά τότε, αυτά που θα πάνε στα γλωσσικά μαθήματα. Γι' αυτό θα χαρώ πολύ κύριε Ναύρατσης αν μπορείτε να μας πείτε λίγα περισσότερα από πού θα αντλήσετε τα κονδύλια για τα πολλά και φιλόδοξα project που μας περιγράψατε. Διότι δεν νομίζω να μας κάνετε ευτυχισμένες εάν τελικά διαπιστώσουμε ότι μας παίρνετε με το ένα χέρι αυτά που μας δίνετε με το άλλο. διότι θα αναγκαστούμε να πούμε σε ανθρώπους που τους έχουμε υποσχεθεί χρηματοδότηση ότι δεν υπάρχουν πλέον λεφτά. Αυτό θα ήταν ε, λίγα ανεσφαλμένο μήνυμα προς τις κοινωνίες μας. Θα χρειαστούν πρόσθετα κονδύλια. Το ερώτημα είναι από πού θα τα βρείτε. Ίσως εκεί να έχετε βέβαια κάποια ευφυή ιδέα που να μπορέσετε να μας κοινοποιήσετε. Και ίσως να τα έχετε ήδη συζητήσει και με τους άλλους επιτρόπους. Ευχαριστούμε. Ε, ο συνάδελφος κ. Λίουερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε κύριε Επίτροπε. Σήμερα το πρωί από τον εισηγητή μας ε, για την ε, έκθεση για το 2020 e ε, πρωτοβουλίε ακούσαμε ότι θα ε, δώσουμε και εμείς μια έκθεση το 2016. Μ' αρέσει λοιπόν που ακούω ότι κύριο σκοπός του πλαισίου αυτού είναι να υποστηρίξει τα κράτη-μέλη. Το επαναλαμβάνω, κύριος στόχος είναι υποστήριξη προς τα κράτη-μέλη για την ανάπτυξη των δικών τους ε, συστημάτων παιδείας και κατάρτισης μέσω ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και αξιοποίησης ε, ε, στοιχείων. Πώς ο κύριος Επίτροπος θα διασφαλίσει ότι θα τηρούνται η επικουρικότητα και οι εθνικές αρμοδιότητες σε αυτόν τον ευαίσθητο τομέα της εκπαίδευσης και θα προσφέρουν επιπλέον αξία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, η κυρία Ευχαριστώ, κύριε Επιτρόπε, για την ομιλία σας. Να ξεκινήσω με ένα γενικό σχόλιο που αφορά τα προγράμματα Creative Europe και Erasmus+. Το έχουμε ξανασυζητήσει πρόσφατα εξακολουθεί ο κόσμος να τα επικρίνει ως υπερβολικά περίπλοκα στην εφαρμογή και νομίζω ότι στην ενδιάμεση αξιολόγηση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου και ελπίζω εκεί να υπάρχει πραγματικά αναθεώρηση και όχι απλά ένα μικρό εγχείρημα να αλλάξουμε την κατάσταση και να τα κάνουμε ευκολότερα γιατί εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα ο κόσμος διαμαρτύρεται ότι τους διώχνουμε από τα ευρωπαϊκά προγράμματα διότι είναι υπερβολικά περίπλοκα δεν έχουν δεν ευχάριστα. Δεν πηγαίνουμε σε αυτά τα προγράμματα και δεν έχει νόημα. Οπότε πρέπει να βρούμε και άλλες δυνατότητες για να προσφέρουμε στου ανθρώπου σε βουλευτική υποστήριξη όταν υποβάλλουν κάποια αίτηση. Τα πράγματα δεν μπορούν να μείνουν όπως έχουν αυτή τη στιγμή. Επίση, θα ήθελα να σχολιάσω ένα από τα πράγματα που είπατε ε, για τον πολιτισμό στην ευρωπαϊκή διπλωματία. Εκεί Είπατε ότι είναι κρίσιμη σημασία όχι απλά η συνεργασία με τι κυβερνήσει, αλλά και η επικοινωνία με πολιτιστικού οργανισμού επιτόπου. Και εγώ θα έλεγα και με μη κυβερνητικέ οργανώσει. Το έχουμε μάθει και από άλλε τέτοιε ε, ε, προσεγγίσεις και από την UNESCO ότι είναι σημαντικό να επικοινωνεί κανείς με τους ανθρώπους επιτόπου, δηλαδή και με τις κοινωνίες των πολιτών. Σας υποστηρίζουμε λοιπόν σε αυτό. Θέλουμε να κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση. Μετά έχω μία ερώτηση Αναφέρατε το ζήτημα του copyright και την ανάγκη εξισορρόπησης της κατάστασης μεταξύ χρηστών και δημιουργών. Θα ήθελα να μου πείτε, επειδή όταν ψηφίσαμε στο Κοινοβούλιο για ε, τη σχετική οδηγία, εκφράστηκε απέτηση από την πλειοψηφία του Κοινοβουλίου η Επιτροπή να απαιτεί κάποιο είδους τέλος ε, από τις εμπορικές πλατφόρμες όταν ε, αξιοποιούν εκεί υλικό που καλύπτεται από κοπήρα. Θέλω να μου πείτε τι έχει κάνει η Κομισιόν σε αυτό το τομέα. Ευχαριστούμε. Εγώ προτείνω να σας δώσω το λόγο να απαντήσετε μετά από τους συντονιστές και μετά θα δώσω το λόγο σε μερικούς άλλους συναδέλφους που ζήτησαν το λόγο. Παρακαλώ κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω με αυτά τα οποία είπατε ότι μία από τις βασικές ευκαιρίες για την οικονομική ανάπτυξη είναι η δημιουργία νέων πόλων παραγωγής και θα πρέπει να βρούμε ένα νέο σύστημα χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες και τις νέες επιχειρήσεις για να μπορούν να ανταγωνίζονται σωστά. Υπάρχει μια συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το αν χρειαζόμαστε ε, μια στρατηγική πλήρως ευρωπαϊκή ή μήπως θα πρέπει να βασιστούμε κυρίως στις βιομηχανίες, στις πολιτικές και στις στρατηγικές των κρατών μελών και απλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσπαθεί να τις βοηθήσει έτσι ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικές. Θα ήθελα και εγώ να πάρω μέρος στη συζήτηση αυτή με νέες ιδέες για την ε, βιομηχανία την ευρωπαϊκή που πρέπει να είναι καινοτόμα. Νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε σημαντικά πλεονεκτήματα και στις ε, ε θα έλεγα τις βιομηχανίες τις σχετικές με την καλλιτεχνική παραγωγή η Ευρώπη είναι πάντα πρωτοπόρος και αν μπορέσουμε να σχεδιάσουμε σωστά χρηματοδοτικά μέσα για την βοήθεια των νεοφιών επιχειρήσεων σε συνεργασία με την αρμόδια επιτροπή, με, την, τον αρμόδιο επίτροπο, τον αντιπρόεδρο Κατάινεν, τον Έτιγκερ και όλους τους σχετικούς επιτρόπους, τότε θα έχουμε νέες δυνατότητες για τη βοήθεια προς τις νέες αυτές επιχειρήσεις. Ελπίζω λοιπόν στο μέλλον να μπορέσουμε να έχουμε κάποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για τη βοήθεια αυτή της ε, δημιουργικής παραγωγής. Υπάρχει λοιπόν μια σωστά συντονισμένη αν θέλετε αντιμετώπιση. Τα προβλήματα με τα μικρά προγράμματα τίθενται πολλές φορές κυρίως από τους Γερμανούς υποψηφίους ότι συγκεντρωνόμαστε πάρα πολύ στα θέματα της πανεπαστημα... ανώτερης εκπαίδευσης και σε μεγάλα προγράμματα. Η απάντηση εδώ είναι ότι λαμβάνουμε εμείς υπόψη μας τις παρατηρήσεις των ίδιων των πολιτών και των εκπροσώπων τους έτσι ώστε το Erasmus Plus να μπορεί να καλύψει και τα τοπικά προγράμματα τα περιορισμένης εμβέλειας. Ήδη από το 2015 ε, πήραμε κάποια μέτρα μείωσης ε, του αριθμού των σχολείων που επιλέγονται, βελτιώνοντας όμως τις δυνατότητες που δίδονται σε αυτά τα σχολεία. Σύμφωνα με κάποια προκαταρκτικά στοιχεία, πάνω από 40% αύξηση των γερμανικών σχολείων το 2015 από ό,τι το 2014. 40% επιπλέον. Ε, το Erasmus Plus για το 2016 η προκήρυξη για, για δηλώσεις ενδιαφέροντος καθορίζει επίσης δύο ε, επίπεδα, καταρχάς τα μικρότερα προγράμματα για την συμμετοχή των μικρών οργανώσεων και των μικρών σχολείων. Θα υπάρξει μια υποδιέρεση δηλαδή για τα προγράμματα μικρής κλίμακας. Και δεύτερον να πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στην Ολομέλεια της Επιτροπής των Περιφερειών και υπήρξε μια ευρυτάτη συνένεση σύμφωνα με το ότι θα πρέπει εμείς να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τις τοπικές οργανώσεις. Θα πρέπει να τις βοηθήσουμε να αναπτύξουν νέα προγράμματα στο πλαίσιο του Erasmus Plus και να τις βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν τη ριζοσπαστικοποίηση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο διότι αυτή είναι η πραγματική αρένα όπου μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη ριζοσπαστικοποίηση. Τα μοντέλα που αναφέραμε μπορούν να βρεθούν εκεί και οι τοπικές αρχές ε, είναι εκείνες που μπορούν να επιτύχουν περισσότερα όσον αφορά την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης. Προσπαθούμε λοιπόν να αναπτύξουμε νέες ε, ευκαιρίες για τις τοπικές ε, ε, αρχές, ε, σχολεία, μικιό ε, τοπικό επίπεδο, αθλητικού συλλόγους για να τους βοηθήσουμε στις προσπάθειες αυτές. Υποστηρίζω ένθερμα την ιδέα του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Το έχω πει επανελειμμένος και σε αυτήν εδώ την Επιτροπή Ωστόσο, η Επιτροπή αποφάσισε να διακόψει προσωρινά οποιαδήποτε πρωτοβουλία για κάποιο ιδιαίτερο ευρωπαϊκό έτος, διότι η Κομισιόν θέλει να προβεί σε μια αξιολόγηση του ρόλου των συνεπειών και της αποτελεσματικότητας ε, των εν λόγω ιδιαίτερων ετών. Ε, υποστηρίζω λοιπόν την ιδέα και αν έχω την ευκαιρία θα εκφραστώ υπέρ ενό ευρωπαϊκού έτου πολιτιστική κληρονομιά, διότι πιστεύω ότι θα προσφέρει τεράστια πλεονεκτήματα για τον τουρισμό, για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, την πολιτιστική διπλωματία, την τοπική ανάπτυξη, την ανάπτυξη πέθρου. υπαίθρου. Είναι μια ολοκληρωμένη ολιστική ευκαιρία, αλλά προς το παρόν θα χρειαστεί να περιμένουμε ε, μέχρι να γίνει η συζήτηση. Αλλά εγώ σίγουρα σε οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση θα υποστηρίξω αυτή την ιδέα του Ευρωπαϊκού Έτου Πολιτική Κληρονομιά. Όσον αφορά το Erasmus Plus, δεν το αποφάσισα εγώ. Είχε αποφασιστεί νωρίτερα να δημιουργηθεί ένα ευρύτερο, πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο με όλα τα προγράμματα, το Leonardo, το Erasmus Plus, το Κοπέρνικο, ώστε να δημιουργηθεί ένα τεράστιο πλαίσιο Erasmus Plus. αλλά και εσείς και όλοι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα προηγούμενα ονόματα που είχαν αυτά τα προγράμματα. Δεν απαγορεύεται. Χρησιμοποιούνται στην καθημερινή, στις καθημερινές συναλλαγές. Ε, συχνά ε, ακούω τα ονόματα Λεωνάρντο Κοπέρνικους. Ε, εάν λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι του βρίσκουν ευκολότερο, μπορείτε φυσικά να χρησιμοποιήσετε τα ονόματα αυτά. εάν είναι έτσι ευκολότερο να προσδιορίσετε τα επιμέρους προγράμματα. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση των νέων υποπρογραμμάτων, έχουμε μια αύξηση στον προπολογισμό του Erasmus ουσιαστικά επιτοπλίστων πρόκειται για νέα χρήματα, νέους πόρους. Σε ορισμένα προγράμματα θα χρειαστεί να επαναπροσανατολίσουμε ή να αναδιαρθρώσουμε τα πράγματα. Ουσιαστικά πρόκειται για το ίδιο ε- ευρύτερο ε, πλαίσιο ερμηνείας. Για παράδειγμα, μαθήματα γλώσσας για μετανάστες, αυτό περιλαμβάνεται στην πολυγλωσσία. Και παλιότερα είχαμε τέτοιους οικονομικούς πόρους, απλά τους αναβαθμίσαμε, ενισχύσαμε ουσιαστικά τους πόρους αυτούς. Πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μεγάλες ανάγκες και τα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών τα χρειάζονται, οπότε αποτελεί βοήθεια, όχι απώλεια. Δεν χάνουμε χρήματα εδώ. Απλά προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα σχολεία εκείνα, τους διδάσκοντες εκείνους και τους μετανάστες πρόσφυγες που πραγματικά βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης. Αυτή είναι μια από τις θεμελιώδεις αποστολές του Erasmus Plus. Το να κάνει την Ευρώπη έναν πιο άνετο χώρο, να ενισχύσει τη συνοχή. Εκεί χρησιμεύει ως μέσο στο να βοηθήσει τη συνοχή της Ευρώπης, της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Η επικουρικότητα με σεβασμό. Ναι, είναι μία από τις θεμελιώδεις μου υποχρεώσεις βάσει των συνθήκων. Δεν μπορώ να παραβιάσω τα όρια της επικουρικότητας. Πολύ απλά. Και όταν προσδιορίζουμε εκείνους στόχους, συχνά, εγώ το πρώτο αυτό μαζί με τους υπουργούς παιδείας, εγώ συχνά περιγραφώ τη δουλειά μου, όχι ως υπερυπουργός παιδείας, αλλά ε, ε, ένας από τους, ότι είμαι ο 29ος υπουργό Παιδείας της Ευρώπης. Ο ρόλος μου είναι να τους διευκολύνω να προσδιορίζουν και να επιτυγχάνουν τους στόχους πολιτικής ε, που έχουν. Αυτός είναι ο χρυσός κανόνας για μένα, το να μην παραβιάζω την αρχή της επικουρικότητας. Και ναι, Συμφωνώ για το ρόλο των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην πολιτιστική διπλωματία. Βρισκόμαστε ε, σύμφωνοι γι' αυτό. Αυτή τη στιγμή συζητάμε και προετοιμάζουμε ε, την οδηγία για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες και την οδηγία για το copyright. και πραγματοποιείται εκτίμηση αντικτύπου αυτή τη στιγμή. Οπότε ε, είναι πολύ νωρί για να πούμε λεπτομέρειε. Ε, οι εργασίε ε, συντονίζονται από τον Αντιπρόεδρο κ. Άντσιπ. Δεν έχουμε ακόμα δει κάποιο λεπτομερές σχέδιο κειμένου, οπότε θα χρειαστεί να περιμένουμε. Ευχαριστούμε και από την κυρία Φεραϊέν και από την κυρία Κάμερεβερτ ε, ζητήθηκε να κάνω μια επιπλέον ερώτηση. Δεν ξέρω αν είναι για αυτό το θέμα, αλλά παρακαλώ. Äh, για το ευρωπαϊκό έτος θέλουμε να δούμε ποια είναι η απήχηση αυτών των ευρωπαϊκών ετών. Από ό,τι θυμούμε γινόταν στο τέλος κάθε έτους μια αξιολόγηση για το ποιε ήταν οι επιπτώσει και θα χρειαζόταν απλά να το διαβάσουμε και τα έχουμε συζητήσει και εδώ αυτά τα πράγματα για παράδειγμα στο έτος του εθελοντισμού ποιε ήταν οι επιπτώσει στις διάφορε χώρε μέλη αυτό ε, δηλαδή, τα χρήματα που δόθηκαν τα κονδύλια που δαπανήθηκαν που, ε, τι απέδωσαν από όσο ξέρω υπάρχουν αυτά τα πράγματα μήπω εκεί οι γενικέ διευθύνσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζουν κάτι Αλλιώς τι να σας πω. Σας εύχομαι πολύ ευχαρίστηση να έχετε όταν θα ψάξετε να βρείτε τα δεδομένα. Και πολλά από τα αίτια αυτά δεν έγιναν καν με ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά από χρηματοδότηση των ίδιων των ενδιαφερόμενων ομάδων. Νομίζω ότι κάποια Ινστιτούτα θα χαρούν πολύ να λάβουν σχετικές μελέτες. Πέτρα Κάμερ Εβερτ. Ευχαριστώ. Ερώτηση για το έρασμο ΣΥΝ. Αν κατάλαβα καλά, κύριε Επιτροπέ, Είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ας το πω αλλιώς, είχαμε αναπτύξει ένα αρκετά περίπλοκο σύστημα σχετικά με την κατανομή των κονδυλίων για τους διάφορους στόχους του προγράμματος. Κατανόησα καλά ότι αυτό που είπατε σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει εξ ιδίων να δαπανίσει αλλού τα χρήματα τα οποία έχουν εγκριθεί και Πού μένει τότε ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σημαίνει δηλαδή ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά βέβαια και το Συμβούλιο Υπουργών, έτσι δεν είναι, ότι εν τέλει θα χρειαστεί να αποφασίσουν εάν τα κονδύλια αυτά θα διατεθούν κάπου αλλού ή εάν θα τροποποιηθεί κάποιο από τα τμήματα του προγράμματος Έρασμος. Μπορείτε να απαντήσετε λοιπόν σε αυτές τις ερωτήσεις και μετά θα δώσουμε το λόγο στους υπόλοιπους συναδέλφους. First, Ως πιστό μέλος της Επιτροπής ε, να σχολιάσω, ευχαριστώ. Για τη δεύτερη ερώτηση. Δεν με τη χρήση των χρημάτων. Αυτή η κοινωνική στόχη προσδιορίζονται μέσα στο Erasmus πλάση η κοινωνική ένταξη, ας πούμε, η ένταξη των νεοαφιχθέντων ε, ανθρώπων, τα μαθήματα γλωσσών ε, εντός της πολυγλωσσίας συμπεριλαμβάνεται. Όλα αυτά έχουν υιοθετηθεί συνενετικά εντός του πλαισίου. Εμείς απλά προβαίνουμε σε μια αναδιάρθρωση εντός αυτών των τομέων, εντός αυτών των δράσεων κλειδιά. Προσπαθούμε δηλαδή να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις που είναι πιστεύω αρκετά σημαντικές αυτήν την εποχή στην Ευρώπη. Δεν είναι ότι δρούμε χωρίς τη συνένεση και τη συγκατάθεση του Κοινοβουλίου. Τους, για τους ίδιους κοινωνικούς στόχους μιλάμε. Απλά χρησιμοποιούμε τα χρήματα. Ουσιαστικά διευρύναμε τη χρήση των χρημάτων βάσει των νέων προκλήσεων. Αλλά συνεχίζουμε όλα τα προγράμματα. Δεν πρόκειται να υπάρξουν περικοπές σε άλλα προγράμματα. Κύριε Επίτροπε, εσείς αναφέρεστε στο ετήσιο σχέδιο εφαρμογής ενός προγράμματος μάλλον το οποίο πράγματι αποτελεί δική σας αρμοδιότητα βάσει της επιτροπολογίας ε, ε, και έτσι θα έχουμε και ένα διάλογο μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Κομισιών ε, με ενημέρωση πριν δηλαδή και μετά τη συνεδρία για το πρόγραμμα, ετήσιο πρόγραμμα θα μεριμνάτε εσείς να μας ενημερώνετε. Έχουμε και την πρώην συνάδελφο ΠΑΚ που ήταν η εισηγήτρια για το Erasmus Plus και τη χαιρετώ. Εμείς τότε είχαμε ορίσει στον κανονισμό για το Erasmus τα κατόφλια, τα, τα ποσοστά ε, για κάθε δράση με ένα ελάχιστο και ένα μέγιστο όριο. Φυσικά κάθε χρόνο πρέπει να επανερμηνεύουμε κάποιες προτεραιότητες, αλλά ο κανονισμός ρητά προβλέπει διακρίσεις, καταμερισμούς του προϋπολογισμού βάσει των στόχων με τρόπο αρκετά ακριβή. Αυτό δεν αποκλείει περιθώριο για κάποιε οριζόντιες στρατηγικέ δράσει, όπω αυτέ που αναφέρατε προηγουμένω αυτή για του μετανάστες για παράδειγμα ε, που αποτελούν κομμάτια ενό νέου θεματολογίου. Κάτι άλλο σημαντικό που εμεί έχουμε ρωτήσει πολλέ φορέ και πολύ ενδιαφερόμενοι το έχουν ζητήσει ε, σε πολλά συνέδρια τα κράτη-μέλη πράγματι μπορούν να εστιάσουν πιο συγκεκριμένες υποκατηγορίες του προγράμματος Εράσμους, στις υποεπικεφαλίδες αλλά βάσει ενό αιτήματο που ακούσαμε, καλό θα ήταν κατά την αναθεώρηση του προγράμματο η λέξη μπορεί να χρησιμοποιήσει ή όχι. Όταν λέει ε, θα πρέπει να αλλάξει σε πρέπει. Ναι, το Erasmus Plus είναι το μεγάλο πλαίσιο, αλλά πρέπει να είναι αναγνωρίσιμα κάποια πράγματα, γιατί αυτό έχει δημιουργήσει σύγχυση. Ε, σε πολλοί κόσμο. Το λέω γιατί μα το έχουν αναφέρει πολλέ φορέ. Λοιπόν, α προχωρήσουμε. Έχουμε τέσσερι συναδέλφου που έχουν ζητήσει το λόγο. Η κυρία Λιμπάσκα, μετά η κυρία Σοντρόβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, πολύ σύντομα πάλι για τον έρασμο. Στη διάρκεια της ακροάσεως που οργανώθηκε από τη δική μας πολιτική ομάδα οι διάφοροι που συμμετείχαν τόνισαν ότι πρέπει ή μάλλον θα πρέπει να μπορούν να συνδέονται οι σπουδές και με μια πρακτική εξάσκηση. Έχετε κάποιες προτάσεις να υποβάλλετε σχετικά εσείς ως Επιτροπή. Δεύτερο, πάλι εδώ μιλώ για τα χρηματοδοτικά. Η ερώτησή μου έχει ως εξής. Δεν μπορούν να βελτιωθούν οι συνέργειες μεταξύ προγραμμάτων όπως για τα πολιτιστικά και για την εκπαίδευση με τα διαρθρωτικά ταμεία και με το επενδυτικό πρόγραμμα Juncker που νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει πηγή χρηματοδοτήσεως και ε, ένα σχόλιο, μάλλον μια παράκληση. Νομίζω ότι πρέπει να αποκαταστήσουμε τον σύνδεσμο μεταξύ πολιτισμού και δημιουργικής βιομηχανίας, δηλαδή creative industry, που νομίζω ότι έχουμε αγνοήσει μέχρι ενό βαθμού. Ιδίως στο, στα πλαίσια του ορίζοντα 2020, διότι σε τομείς όπως ο πολιτισμός, και στην παιδεία. Η creative industry μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Μπορείτε να κάνετε κάποια, να ασκήσετε κάποια πίεση, να κάνετε κάποιο λόμπι, ώστε να αναπτυχθούν περισσότερες συνέργειες μέσα στο πλαίσιο αυτό για τον ορίζοντα 2020. Ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη συνάδελφος. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Εκτιμώ το πρόγραμμα εργασίας σας και τις κατευθύνσεις τις οποίες είπατε ότι θα ακολουθήσετε. Θα ήθελα και εγώ να επιβεβαιώσω προς τους συναδέλφους ότι το Εράσμος λειτουργεί πια με ανοιχτό και επικοινωνιακό τρόπο και ανταποκρίνεται όταν ζητάμε αλλαγές για συγκεκριμένες κοινότητες, για συγκεκριμένες ομάδες παιδιών και ομάδες διδασκόντων απαιτούνται μερικές φορές να υπάρχουν αλλαγές στις διαδικασίες. Υπάρχει η δυνατότητα πάντως για να το πετύχουμε αυτό. Ζούμε σε δύσκολες εποχές. Είπε ο κύριος Τίμερμανς ότι αντιμετωπίζουμε την ισχυρότερη κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη στιγμή που δημιουργήθηκε. Συνεπώς λοιπόν η σημασία της εκπαίδευσης είναι πολύ μεγάλη, ιδιαίτερα αυτή την εποχή. Εμείς οι πολιτικοί αντιμετωπίζουμε πολλές προκλήσεις και στον τομέα τον κοινωνικό και στον τομέα της ασφάλειας προσπαθούμε να συζητήσουμε νέες απαντήσεις και να βρούμε τον τρόπο να ανταποκριθούμε στις ευθύνες μας. Οι ερωτήσεις τίθενται από φοιτητέ, από μαθητές, από διδάσκοντες, αντιμετωπίζουν προβλήματα σε καθημερινή βάση στην Τσεχία προετοιμάζω ένα, ένα, μια στρογγύλη τράπεζα για δασκάλους και καθηγητές έτσι ώστε να ενημερώνονται σωστά για τις αποφάσεις των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. γιατί δεν έχουν τις σωστές πληροφορίες, τις αντικειμενικές πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά λοιπόν για την πληροφόρηση και την στήριξη μεθοδολογικά. Θα ήθελα να υπάρχουν κάποια μέσα ενημέρωσης σε κοινοτικό επίπεδο για τα Υπουργεία Παιδείας σε οριζόντιο επίπεδο, ενώ ότι τα Υπουργεία Παιδείας πολλές φορές δεν γνωρίζουν πλήρως τις δυνατότητες που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν οι προσπάθειες των Εθνικών Υπουργείων να παρακολουθούνται σωστά και νομίζω ότι αυτό θα δώσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια πραγματική εικόνα και πρέπει να βρούμε και τα σωστά επιχειρήματα βέβαια τα οποία να χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις εθνικές υπηρεσίες. όταν λαμβάνονται κάποιες αποφάσεις για επιμέρους περιπτώσεις σε εθνικό επίπεδο. Ποιος είναι ο υπεύθυνος για να παρακολουθήσει την πραγμάτωση αυτής της απόφασης. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας και μιας εκπαιδευτικής δράσης. Ποιος θα είναι υπεύθυνο λοιπόν, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Ε, πρώτα η Word και μετά ο κύριος Γραμματικάκης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ τον Επίτροπο για τα καλά του λόγια, για την έκθεσή μου για τον διαπολιτισμικό διάλογο. Είμαι ικανοποιημένη νομίζω από το αποτέλεσμα. Είχα θετική ανταπόκριση από εκπαιδευτές, από δασκάλους, καθηγητές, οργανώσεις που ελπίζω θα χρησιμοποιήσουν την έκθεση έτσι ώστε να αποκτήσουν περισσότερη εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους και να αποκαταστήσουν τον διάλογο ανάμεσα στις διαφορετικές κατηγορίες. Να σημειώσω επίσης ότι συμφωνώ με πολλά από αυτά τα οποία ακούσαμε εδώ για την επιχειρηματικότητα. Ίσως θα πρέπει να βάλετε και το επίθετο κοινωνική επιχειρηματικότητα. Να μην μιλάμε αποκλειστικά για την επιχειρηματικότητα αυτή καθεαυτή που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πρακτικές οι οποίες είναι καταχρηστικές. Ε, ε, πολλές φορές ε, η επιχειρηματικότητα και οι επιχειρήσεις είναι κάτι το θετικό, αλλά υπάρχει και η κοινωνική επιχειρηματικότητα την οποία οι νέοι κατανοούν πολλές φορές εύκολα γιατί πιστεύουν ότι μπορεί να προσφέρει, προκαλεί το ενδιαφέρον τους και πολλές φορές υπάρχουν προγράμματα ήδη στα διάφορα σχολεία σχετικά με το δίκαιο εμπόριο, το fair trade. Κάτι άλλο το οποίο έχει επίσης μεγάλη σημασία είναι το λεγόμενο STEM και όχι STEM, δηλαδή πρέπει να μην ξεχνάμε τις δυνατότητες που παρέχουν οι ανθρωπιστικές σπουδές. Εμείς στο Μάντσεστερ που είναι μια τεράστια πόλη έχουμε μια μεγάλη συνάντηση τον Ιούλιο ε, για ε, την ε, βιομηχανία και έχουμε ένα μεγάλο κεφάλαιο της συνάντησης για τη σχέση βιομηχανίας και πολιτισμού και όπως έχω ήδη πει θα υπάρξει μια μεγάλη συνάντηση και με τον Γενικό Διευθυντή της Siemens και μαζί θα προσπαθήσουμε ε, να βοηθήσουμε τη Siemens να κατανοήσει ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Um, um, uh, Σχετικά τώρα με τις βέλτιστες πρακτικές. Αυτό είναι κάτι το οποίο διαπερνά θα έλεγα πάρα πολλά επιμέρους θέματα. Ξέρω ότι μαζί 28 χώρες μέλη δημιουργούν τεράστιες δυνατότητες στον τομέα του διαμοιρασμού των βέλτιστων πρακτικών. Αυτό είναι βασική ε, προστιθέμενη αξία. Είναι κάτι το οποίο λειτουργεί πολλαπλά και αμφίδρομα Ξέρουμε ότι πολλά γίνονται σε πολλές χώρες με πολύ ενδιαφέρον για θέματα όπως η κατάρτιση ε, των ε, αυτών που καταρτίζουν με τη σειρά τους, η εκπαίδευση των εκπαιδευτών σαν παράδειγμα και πολλά μένει να προσφέρουμε ακόμα ο ένας τον άλλο. Και πάρα πολύ μεγάλη σημασία επίσης έχουν και οι ατυπικές διαδικασίες εκπαίδευσης. Συγγνώμη αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο λέει η Πρόεδρος. Ο κύριος Γραμματικάκης. Εγώ θα είμαι πολύ σύντομος κύριε Επίτροπε ως συνήθως ε, πρώτα απ' όλα με κάτι που φαίνεται ότι δεν σχετίζεται με τα σημερινά αλλά σχετίζεται πάρα πολύ. Η κυρία Πρόεδρος είχε την καλοσύνη να το αναφέρει το πρωί. Να σας πληροφορήσω λοιπόν και ως καθηγητή του, αν θυμάμαι καλά, της πολιτικής επιστήμης, το οποίο σας θυμά ιδιαίτερα, ότι φέτος εορτάζονται στη Θεσσαλονίκη σε ένα παγκόσμιο συνέδριο τα 2.400 χρόνια από τη γέννηση του Αριστοτέλη ενός εκ των σπουδαιότερων βέβαια φιλοσόφων, πολιτικών φιλοσόφων, επιστημόνων και γενικών ιδρυτή της σημερινής ευρωπαϊκής σκέψης. Το λέω αυτό σαν μια πρόσκληση και προς εσάς, όπως απίφθηνα και την απεδέχτη κυρία, στην κυρία Κώστα και σε κάθε ένα παριστάμενο εδώ από τους αγαπητούς συναδέλφους, το συνέδριο έχει υιοθετηθεί από την UNESCO ήδη. Έχει ήδη 600 παγκόσμιες συμμετοχές. Παρακαλώ προσέξτε το. Και είναι λυπηρό μετά από αυτό που κάνει μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα με τόση μεγάλη συμπαράσταση να ακούω ότι τίθεται ακόμα σε συζήτηση το έτος της πολιτιστικής κληρονομιάς. Έλεος. Έλεος. Το αυτονόητο συζητάμε κύριε Επίτροπε και χαίρομαι που τουλάχιστον εσείς έτσι μας είπατε υποστηρίζετε πάρα πολύ αυτή την ιδέα. Πολύ κουβέντα έγινε σήμερα και κλείνω για το έρασμος. Θετική, αρνητική, άκουσα πάρα πολλά. Θα σας δώσω μια πληροφορία γιατί από κάπου αναφέρθηκε ότι πιθανόν δεν υπάρχει ένας απόλυτος συντονισμός. Στην πατρίδα μου που ζει υπό οδυνή κρίση, την πατρίδα του Αριστοτέλη και άλλων φιλοσόφων και μου προσωπικός που δεν τους φτάνουν ούτε στον νυχάκι τους, αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα έρασμους έχει να, να λειτουργήσει από το 2014. Παρακαλώ. Φαντάζομαι να σας ενημέρωσε το γραφείο σας ή να υπάρχει μια επικοινωνία με το Υπουργείο της Ελλάδος. Ε, το 2014 δεν έχουν πληρωθεί οι άνθρωποι, το 2015 δεν προκυρήθηκε καθόλου και το 2016 ήρθε κάποια μυστήρια εντολή για αναστολή του προγράμματος. Αυτά τα στοιχεία τα έχω παραδώσει και στην πρόοδο της Επιτροπής. Ευχαρίστω να σας τα στείλω και εσάς. Οι φοιτητέ, οι νέοι άνθρωποι είναι απεγνωσμένοι και κλείνω με το ότι δεν, αν θέλετε, με ανησύσε και η δική σας κατά κάποιο τρόπο απολύτως κατανοητή έτσι, συνένεση με το ένα μέρος των κλασικών χρημάτων του έρασμου, έτσι το κατάλαβα εγώ, με αναδιάρθρωση, μετακίνηση και εν περιπτώσει λόγω των απίστευτων πιέσεων που αυτή τη στιγμή ζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πιθανό να πάνε σε άλλες κατευθύνσεις. Έτσι το ερμήνευσα, ελπίζω να μου το διαψεύσετε. Ευχαριστούμε. Πέτρα, είπατε ότι θέλετε ένα follow-up και μετά να κλείσουμε την απάντηση. Ευχαριστώ που μου δίνετε πάλι το λόγο. Μένω κατά κάποιο τρόπο άναυδη, ας το πω έτσι. Επανέρχομαι στο έρασμο Συν, διότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματικά το έχουμε κλείσει στην καρδιά μας και θα τα πω λίγο πιο σαφώς. Ίσως κύριε Ναύρατσιτς να ακούτε τώρα τα οργισμένα μας λόγια ενώ δεν ευθύνεστε εσείς αλλά η προηγούμενη επιτροπή να μην... Ε, δεν έχουμε όμως μόνο απλώς την εντύπωση σχετικά με τα όσα ακούμε για την εφαρμογή του προγράμματος, ότι δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές διατάξεις που δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που έχουμε αποφασίσει εμείς. Και τώρα φαίνεται να προστίθεται από πάνω και το ότι τα όσα έχουμε ήδη αποφασίσει ερμηνεύονται με τέτοιον τρόπο ώστε να προσαρμόζονται στην υφιστάμενη κατάσταση. Παράδειγμα, λέμε κάτι εκεί για την προώθηση της πολυγλωσσίας στο πρόγραμμα. Ναι βεβαίως πάντα το θέλαμε αυτό να υπάρχει το στοιχείο. Όμως προώθηση της πολυγλωσσίας κατά τη δική μου κατανόηση δεν σημαίνει προώθηση ή χρηματοδότηση γλωσσικών ε, προγραμμάτων για πρόσφυγες. Δεν σημαίνει αυτό. Εάν τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα στην ανάγκη προσπαθεί αυτά που έχουμε περιγράψει εμείς ως στόχους να τα τεντώσει τόσο πολύ ώστε να μην έχουν πια καμιά σχέση σχεδόν με αυτά που είχαμε αρχικώς εκφράσει εμείς ως πρόθεση αναμένω τουλάχιστον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφόσον προγραμματίζει τέτοια πράγματα τουλάχιστον να μιλήσει με εμάς ειλικρινώς και να μας ρωτήσει εάν μπορούμε να συμφωνήσουμε εάν μέσα στις εξελισσόμενες αυτές καταστάσεις όπου βρισκόμαστε μπορούμε και να συμφωνήσουμε και αν όντω αυτά που κάνει ανταποκρίνονται στην ε, εκπεφρασμένη πολιτική μας βούληση. Γνωρίζουμε ότι τα χρήματα είναι πολύ περιορισμένα. Γνωρίζουμε ότι τα χρήματα απορροφώνται και απολύτως. Εάν τώρα διαρκώς από αυτά τα ε, ελάχιστα χρήματα του έρασμος καλούμαστε να χρηματοδοτήσουμε και πράγματα που δεν εννοούσαμε όταν αποφασίσαμε αυτά που αποφασίσαμε. Αναμένω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσέλθει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μιλήσει μαζί μα και να προ... κοιτάξει να συμφωνήσει μαζί μα. Και η επανεξέταση review που θα έχουμε μπροστά μα αποτελεί την κατάλληλη ευκαιρία. Σα παρακαλώ λοιπόν από καρδιά την έκκληση αυτή που σα απευθύνω να την ακούσετε, να την εισακούσετε και να ανταποκριθείτε. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να διευκρινιστεί και πάνω σε αυτό νομίζω Επίτροπε θα πρέπει να υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες ε, σε μια άλλη αφορμή συνάντησης. Να θυμίσω εδώ ή μάλλον Βέντα πρώτα και μετά θα ήθελα να κάνω εγώ κάποιες παρατηρήσεις. Βέντα. Συνειδητοποιώ ότι τέθηκαν πάρα πολλές ερωτήσεις και αρκετά δύσκολες ερωτήσεις και γι' αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις απαντήσεις σας. Μιλήσατε και για τον αθλητισμό. Ο αθλητισμός είναι κάτι το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την καλύτερη κοινωνική απορρόφηση των μεταναστών και των προσφύγων. Ήταν ενδιαφέροντα αυτά που είπατε για, τους, ε, για την ε, αθλητική διπλωματία. Ε, ο αθλητισμός σαν καρπός αλλά και παράγον της κοινωνικής συνοχής έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία πέρα από τις ίδιες τις αθλητικές επιδόσεις. Αναφερθήκατε επίσης στην FIFA και σε άλλες οργανώσεις ευρωπαϊκές ημί. Πέραν της αυτονομίας αυτών των οργανώσεων πέρα από διάφορους μάνατζερ οι οποίοι πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι αυτοί επιθυμούν. Αναφερθήκατε και σε διάφορα σκάνδαλα με ε, ουσίες και τα λοιπά. Είναι απλά οικονομικό το θέμα, ε, δεν ξέρω πού μπορείτε να παρέμβετε. Τι μέσα λοιπόν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κύριε Επίτροπε έτσι ώστε να υποχρεώσουμε αυτές τις μεγάλες αθλητικές οργανώσεις να συνεργαστούν μαζί μας έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες τους με σωστότερο τρόπο. Όχι μόνο για να τις διαφημίσουμε αυτές τις οργανώσεις αλλά να συμφωνήσουν και αυτές να βοηθήσουν σε μεγάλα θέματα κοινωνικά όπως η απορρόφηση των μεταναστών. Ξέρετε ότι υπάρχει μια διοργανική ομάδα που συνεργάζεται και με τη FIFA και νομίζω ότι οι οργανώσεις αυτές όπως η FIFA έχουν πάρα πολλά χρήματα και θα μπορούσαν να βοηθήσουν έτσι ώστε να οργανώσουμε με διαφορετικό τόπο τις πρωτοβουλίες μας. κάποιες σύντομες σκέψεις. Νομίζω ότι η συζήτηση που προηγήθηκε ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Εκτιμήσαμε δεόντως, κύριε Επίτροπε, τις λεπτομέρειες και το βάθος το οποίο αναφερθήκατε σε αυτές. Πρέπει να υπάρχει, όπως είπατε, συνεργασία ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μέχρι τώρα φαίνεται και ελπίζω να αλλάξουν τα πράγματα γιατί όσο περισσότερη εκπαίδευση υπάρχει τόσο περισσότερη παιδεία και η Ευρώπη αυτή τη στιγμή κινδυνεύει γιατί στον τομέα του πολιτισμού και στον τομέα της εκπαίδευσης τα πράγματα υποτιμήθηκαν. Πρέπει λοιπόν και στα πλαίσια της Επιτροπής Γιούνκερ να πούμε ότι τα πράγματα λειτουργούν με οικονομικίστικο σε εισαγωγικά βλέμμα. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια διαφορετική κουλτούρα που θα βοηθήσει την Ευρώπη να γίνει πιο ανθεκτική και τους κατοίκους της Ευρώπης, τους πολίτες της Ευρώπης να νιώσουν πιο άνετα μέσα σε αυτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ουσία θα έλεγα συνδυάζεται με άλλα 28 εθνικά συστήματα παιδείας τα εθνικά συστήματα παιδείας φυσικά είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών και σε οργανωτικό επίπεδο και σε επίπεδο επιλογής της διδακτέας ύλης. Αλλά ο στόχος μας είναι με περισσότερο φιλόδοξος να δημιουργήσουμε έναν ευρωπαϊκό χώρο πολιτισμού και έρευνας και να επιτρέψουμε μέσω της αμοιβαίας αναγνώρισης των συστημάτων, της αναγνώρισης των τίτλων, και με τις συστάσεις επίσης τις οποίες κάνετε εσείς ε, στα διάφορα κράτη-μέλη ε, για την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού. Να βελτιώσουμε τις δυνατότητες έτσι ώστε όλοι οι νέοι και όχι μόνο οι νέοι να νιώσουν Ευρωπαίοι πολίτες, να υπάρχει δηλαδή ε, δικαιοσύνη στην αμοιβαία αναγνώριση, να δημιουργηθούν δίκτυα αμοιβαίας αναγνώρισης όπως είπα και ένα δεύτερο σημείο τώρα για τη βιομηχανία και την παραγωγή πνευματικών έργων κτλ. Ε, μου αρέσει που δίνετε σημασία σε αυτό και θα περιμένουμε η Επιτροπή μας τις προτάσεις σας ε, μετά από τις τελευταίες αποφάσεις οι οποίες πρόσφατα ελήφθησαν μετά την Πράσινη Βίβλο και τη δική μας έκθεση δεν ακούσαμε και πάρα πολλά από πλευρά της Επιτροπής. Δεν υπήρξε μια κατευθυντήρια θα έλεγα τάση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Γι' αυτό αφορά και τη Γενική Διεύθυνση Πολιτισμού και τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων. Λοιπόν, είναι ο τομέας μας αυτός ανταγωνιστικός όχι σαν αγορά μόνο αλλά κυρίως σαν, ε, σε επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης. Το πακέτο skills λοιπόν, ικανότητες, θα πρέπει να μην αγνοήσει τον πολιτισμό, την πολιτιστική κληρονομιά, τις εκδόσεις, τη μουσική, τα ραδιοτηλεοπτικά γιατί όταν μιλάμε για τον πολιτισμό, μιλάμε γενικά για τον πολιτισμό, λες και ήταν κάτι το δευτερεύον χωρίς να διευκρινίζουμε το περιεχόμενό του. Και να μην ξεχνάμε ότι είναι ένας νέος τομέας ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. Αντιπροσωπεύει πάνω από το 5% του ΑΕΠ ο τομέας αυτός. Είναι στρατηγική σημασίας και η απασχολησιμότητα των νέων κυρίως είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει πολύ. Ένα τελευταίο σημείο για την πολιτιστική κληρονομιά. Ασκήθηκε κριτική στο ότι η Επιτροπή γενικότερα επανέρχεται στο θέμα αυτό και τελικά το 2016 δεν ξέρουμε τι χρονιά είναι, δεν ξέρουμε τι, δεν υπάρχει δηλαδή μια συγκεκριμένη προσπάθεια που να γίνεται, υπάρχει μια κάποια αδράνεια. Δεν κατηγορώ εσάς τον ίδιο προσωπικά. Βλέπουμε όμως τι γίνεται τα προηγούμενα, τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Το Συμβούλιο Υπουργών Πολιτισμού εκφράστηκε επίσημα υπέρ της Ευρωπαϊκής Χρονιάς Πολιτισμού το Δεκέμβριο του 2015 με Ιταλική Προεδρία. Είχα πάει στη Ρώμη χθε σε μια πρωτοβουλία με τον Υπουργό Πολιτισμού και ε, μου έστειλαν υπουργοί, είπε κάποιοι υπουργοί από την Γερμανία, από την Ιταλία από τη Γαλλία και από το Λουξεμβούργο όπου είπαν ότι το, Συμβούλιο ενδιαφέρεται γι' αυτό, εκφραστήκαμε και εμείς υπέρ φυσικά επίσημα, με μεγάλη πλειοψηφία για την πολιτιστική κληρονομιά. Έχετε λοιπόν τα μέσα για να προωθήσετε το θέμα αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί νομίζω ότι το να εγκαταλείψει κανείς αυτή την προοπτική η οποία ζητήθηκε από πολλούς φορείς στην Ευρώπη όπως τα Europa Nostra. Ε, νομίζω λοιπόν ότι αυτό θα ήταν πολιτικό λάθος. Και μια τελευταία παρατήρηση, το θέμα της χρηματοδότησης. Στέχθηκαν επιπλέον θέματα για τη χρηματοδότηση. Έφτασε η στιγμή στα πλαίσια της οποίας και δεν αναφέρομαι μόνο στα συγκεκριμένα θέματα της χρηματοδότησης όπου θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας στείλει μια επιστολή για τους επιπλέον πόρους για το Εράσμους. Κάτι το γενικότερο. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε δύο καινοτομίε το 2016. Η πρώτη ονομάζεται νέο χρηματοδοτικό μέσο για την δημιουργική Ευρώπη, πολιτισμός, τηλεόραση, κινηματογράφος κτλ καθυστερήσαμε σε επίπεδο τεχνικό. Τώρα ξεκινάει αυτό το μέσο, είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο και νομίζω ότι και η Γενική Διεύθυνση Connect ε, και η δική σας νομίζω ότι το θέμα αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για όλους. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς να ακολουθήσουμε μια διαφορετική πορεία στον τομέα αυτό, μιας και συζητιέται σε επίπεδο διαφόρων γενικών διευθύνσεων. Το, το αυτό το Ταμείο για τις Στρατηγικές Επενδύσεις, το οποίο μέχρι τώρα δεν έχει στείλει ούτε ένα ευρώ στα εκτελεστικά, στα προγράμματα του πολιτισμού, γιατί θεωρούνται πιο επικίνδυνα και λιγότερο ελκυστικά γιατί να μην συνδυαστούν όλα αυτά τα όλες αυτές οι χρηματοδοτικές ροές σε μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα συγκέντρωσης των πόρων έτσι ώστε να δώσουμε διαφορετικές δυνατότητες και στους επενδυτές και στα πιστοτικά ιδρύματα και στους stakeholders γενικά και να καταστήσουμε τα προγράμματα αυτά ελκυστικά και σε εθνικό επίπεδο. Ξέρω ότι τα θέματα αυτά γίνονται, ε, είναι σε συζήτηση ανάμεσα στις διάφορες γενικές διευθύνσεις. Είναι ένα θέμα το οποίο ε, θα έλεγα αφορά όλες τις, ε, όλους μας. Πρέπει να βρούμε επιπλέον πόρους γιατί αλλιώς ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ υψηλός. Και τελειώνω τώρα για την εκπαίδευση των μεταναστών. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ε, φυσικά και πρέπει να υπάρξουν εγκάρσιες δράσεις του Εράσμου τα οποία ανακαλύπτουν τομείς όπως η δημιουργική Ευρώπη κτλ. Και να προσφέρουμε στους μετανάστες και τις πολιτιστικές αυτές ομάδες και συλλόγους δυνατότητες έκφρασης. Είναι μια στοχευμένη αν θέλετε κατηγορία. Θα πρέπει όμως να βρεθούν συμπληρωματικοί πόροι μετά από Παρίσι, οι αποφάσεις που λαμβάνονται σημαίνουν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει κάποιες από τις προτεραιότητές της. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει απλό θέμα αδράνειας. Οι πολιτικές δεν ανταποκρίνονται με τα προγράμματα. Τα προγράμματα αποφασίζονται και οι πολιτικές πρέπει να εφαρμόζονται με τις απαραίτητες καλύψεις σε επίπεδο δημοσιονομικό από το Μογκερίνι μέχρι το Γιούνκερ όλοι λένε ότι χωρίς πολιτισμό, χωρίς επενδύσεις δεν υπάρχει εξωτερική πολιτική, δεν υπάρχει πολιτική γειτονία, δεν υπάρχει πολιτική μετανάστευσης, δεν υπάρχει πολιτική ασφάλειας. Και όμως δεν γίνεται τίποτα σε επίπεδο χρηματοδότησης. Αυτό είναι απαράδεκτο. Πρέπει να είμαστε πιο απαιτητικοί και να προσπαθήσουμε να διευκρινίσουμε ότι θα σας βοηθήσουμε όταν ζητήσετε περισσότερους πόρους. Και το θέμα δεν είναι να παίρνετε την μπουκιά από το στόμα, από τα παιδιά του Εράσμου τα οποία με ελάχιστες υποτροφίες προσπαθούν όπως να καλύψουν τις ανάγκες τους. Θα πρέπει να υπάρξει ικανοποιητική χρηματοδοτική κάλυψη. Ένα το πετύχαμε. Προσπαθήσαμε να αυξήσουμε στα πλαίσια της ανθρωπιστικής βοήθειας Προσπαθήσαμε με την έκθεση του Κοινοβουλίου και με μια θετική τελικά απάντηση από πλευράς του Επιτρόπου για την ανθρωπιστική βοήθεια 27 εκατομμύρια να δοθούν επιπλέον το 2017 για την αύξηση της ποσόστοσης που έχει σαν στόχο την εκπαίδευση ε, στους, στα στρατόπεδα των προσφύγων ή στους οικισμούς των προσφύγων για τα παιδιά που είναι σε κατάσταση ανάγκης. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το μέσο αυτό γιατί αυτό το οποίο πηγαίνει στην εκπαίδευση είναι το 2% της ανθρωπιστικής βοήθειας και έτσι θα αποφύγουμε τη ριζοσπαστικοποίηση. Υπάρχουν 100.000 παιδιά στην Τουρκία για τα οποία παρέχονται υποτίθεται κάποιες υπηρεσίες. Είναι περίπλοκο το θέμα, σας τα λέω όλα κάπως σχήμα, αλλά εν πάση παθιάζομαι γι' αυτά. Είναι θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν όλους. Άκουσα με ικανοποίηση τα νέα θέματα τα οποία θέσατε και νομίζω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε, να θεωρήσουμε ένα τον άλλο σύμμαχο και να μην κάνουμε φτωχότερα όμως τα προγράμματα που ήδη έχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, να πω κάτι για τις παρατηρήσεις της κυρίας Κάμερβερτ. Όταν αλλάζουμε το σημείο εστίασης, νέα σημεία εστίασης, ε, όλα αυτά γίνονται εντό του πλαισίου ευελιξίας και συνήθως γίνεται και κάποιος διάλογος με την Επιτροπή, οι υπηρεσίες μου, το γραφείο μου, όλοι μας βρισκόμαστε σε ε, μόνιμη επαφή σας, διατηρούμε ενήμερους. Η επόμενη τέτοια εκδήλωση θα είναι στην ε, ε, συνάντηση της Επιτροπής τον Απρίλιο. Κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε καλύτερο για να σας διατηρούμε ενήμερος σε σχέση με τις τελευταίες εξελίξεις και προτεραιότητες και τα σημεία εστίασης. Ε, κυρία Λιμπάτσκα, για την ερώτησή σας, αν κατάλαβα καλά, Αναφερθήκατε στις μαθητείες και στο συνδυασμό επαγγελματικής κατάρτισης και προγραμμάτων Erasmus+. Έχουμε ένα υποπρόγραμμα εντός του Erasmus+, το οποίο υποστηρίζει τα προγράμματα μαθητείας, περίπου 50.000 ε, προγράμματα μαθητείας ετησίως υποστηρίζονται μέσω αυτού. Κοιτάξτε, δεν καταλαβαίνω. Ε, εν συντομία, κύριε Επίτροπε, να σα κάνω μια ερώτηση. Εάν κάποιος φοιτητή φύγει με εράσμου σε μια άλλη χώρα, μπορεί καθώς φυτά να κάνει και κάποιο, ε, ε, ε, ε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, κάποιο, κάποια πρακτική εξάσκηση. Eh, you paid by, eh, Που να αμείβεται από κάποιον άλλο ή από το πρόγραμμα. Ε, χωρίς μικρόφωνο δυστυχώς μιλάει η κυρία. Χωρίς χωρίς μικρόφωνο. Συγγνώμη λέει η κυρία Λιμπάτσικα. κυρια λιμπατσικα ενω αυτός ο οποίος υποδέχεται τον σπουδαστή ο φορέας που θα υποδεχθεί τον σπουδαστή να πληρώσει κιόλα. Αλλά κυρίως να μην υπάρξει σύγκρουση ανάμεσα στον κύκλο των μαθημάτων και στην δυνατότητα ολοκλήρωσης της πρακτικής εξάσκησης. Αυτός που θα πληρώσει θα είναι η επιχείρηση η οποία θα υποδεχτεί τον σπουδαστή και θα του προσφέρει το, την πρακτική εξάσκηση. Θα μπορούσατε να το διευκρινίσετε αυτό ενδεχομένως ε, με κάπως καλύτερη ενημέρωση για τους πόρους του Εράσμους ε, φέτος ε, για αυτές τις πτυχές. Όταν θα μα κάνετε λοιπόν αυτή την ενημέρωση μπορείτε να διευκρινίσετε και αυτό ενδεχομένως και να απαντήσετε στην ερώτηση αυτή. Ωραία. Thank you. <coughs> Uh, discuss, agenda Uh, ουσιαστικά ε, ε, το θεματολόγιο αυτό είναι μια στρατηγική. Σχεδιάζει κατευθύνσεις για την επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση, τα εκπαιδευτικά συστήματα, την αγορά εργασίας και για πιο ευέλικτα τμήματα της εκπαίδευσης. Η υλοποίηση του θεματολογίου για τις δεξιότητες αποτελεί ουσιαστικά καθήκον των κρατών μελών όπως και η εγγύηση για τους νέους, όπως σχεδόν ε, όλες όλα τα μέσα και εργαλεία για τις πολιτικές απασχόλησης εναπόκειται στα κράτη-μέλη το πόσο αποτελεσματικοί θα είμαστε στην εφαρμογή. Εμείς φυσικά μπορούμε να αφιερώσουμε προγράμματα για να τα βοηθήσουμε ευαισθητοποιώντας τον κόσμο για το θέμα των δεξιοτήτων αλλά ουσιαστικά τα κράτη-μέλη είναι αυτά που ε, έχουν την ευθύνη της ε, υλοποίησης των προγραμμάτων. Συμφωνώ απόλυτα με την Τζολι Βόρτ για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, αν και έφυγε. Α, εδώ βρίσκεται. Ε, και μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις πιστεύω θα είναι η χρήση και η εκμετάλλευση των ευκαιριών στον τομέα της άτυπης εκπαίδευσης διότι για την κοινωνική συνοχή η άτυπη εκπαίδευση είναι ο πιο ευέλικτος τρόπος ένταξης των αφιχθέντων ανθρώπων είτε σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, είτε σε πολιτιστικές δραστηριότητες, είτε σε αθλητικές δραστηριότητες. Η άτυπη εκπαίδευση προσφέρει πολλές καλές ευκαιρίες που μπορούν να αξιοποιηθούν για την κοινωνική ένταξη. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση για ε, την επέτειο της γέννησης του Αριστοτέλη. Δεν θα έλεγα ότι η Ελλάδα είναι μικρή χώρα. Ξέρετε, δεν είναι μόνο θέμα έκτασης ή πληθυσμού. Η πολιτιστική κληρονομιά είναι τεράστια και φυσικά και η πολιτική ιστορία μιας χώρας σαν την Ελλάδα είναι τεράστια. Και εξού και ο πλούτος της. Πρέπει να πω ότι είναι οδυνηρό το ότι υπάρχουν προβλήματα με το Erasmus Plus ε, στην Ελλάδα. Από όσο ξέρω, ουσιαστικά οι εθνικοί φορείς ε, είναι που αντιμετωπίζουν προβλήματα στο θέμα αυτό. Είμαστε σε στενή επικοινωνία με τις ελληνικές αρχές και ελπίζω να μπορέσουμε να διευθετήσουμε το πρόβλημα και να επανεκκινηθεί το όλο πρόγραμμα Erasmus στην Ελλάδα γιατί ήσασταν πολύ δραστήριοι σε αυτό το πρόγραμμα παλιότερα, οπότε ελπίζω να διορθωθεί η κατάσταση. Για τον αθλητισμό τώρα, συμφωνώ με το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο αθλητισμός ε, ε, στην αθλητική διπλωματία. Όπως μόλι ανέφερα, έχουμε μια ομάδα εργασίας υψηλού επίπεδου, η οποία διερευνά τι ευκαιρίε που θα μπορούσε να προσφέρει η αθλητική διπλωματία. Έχουμε πολλά θετικά παραδείγματα ε, κοινωνικής ένταξης ε, χάρη στον αθλητισμό στις 2 Μαρτίου με την ε, Sports Intergroup Group θα πάμε εδώ στο Κράινεμ στο αθλητικό κέντρο του Κράινεμ όπου τρέχει ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης και έχουμε πολλά ε, ικανοποιητικά παραδείγματα σε διάφορα μέρη ε, από τον Brussels Sports ε, που βοηθούν για την ένταξη των Ρωμά, των μειονοτήτων, των προσφύγων. Μπορούμε λοιπόν να βασιστούμε σε αυτά τα παραδείγματα και να τα αξιοποιήσουμε ως καλά μοντέλα για τη μελλοντική συνεργασία. Έχουμε και μια άλλη ομάδα εργασία ε, για τη χρηστή διακυβέρνηση στον τομέα του αθλητισμού. Αυτή τη στιγμή αυτή είναι η κύρια πλατφόρμα ε, συνεργασία με του μεγάλου αυτού αθλητικού οργανισμού. Οι εκπροσωποί τους ε, συμμετέχουν στις δραστηριότητες της εν λόγω ομάδας εργασίας. Αποτελέσματα θα έχουμε μέχρι το καλοκαίρι ελπίζω. Και οι αθλητικοί οργανισμοί είναι εκείνοι που θα αποφασίσουν κατά πώς θα συμβάλλουν ενεργά στην υλοποίηση των αρχών χρηστής διακυβέρνησης και κατά πόσο θα βοηθήσουν να βελτιωθούν τα στάνταρ για τον αθλητισμό και το περιβάλλον σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την επίσκεψη αυτή, η οποία ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, εκδηλώθηκε έντονο ενδιαφέρον από τους συναδέλφους. Όπως βλέπετε Μας αρέσει που στρέφεται η προσοχή όλης της Επιτροπής σε αυτές τις στρατηγικής σημασίας κατά με προτεραιότητες ε, που θα ενισχύσουν την αισθή ηθαγένειας και ταυτότητας. Να υπενθυμίσω ότι φέτος ε, είναι 20η επέτειος ε, του σχεδίου του προγράμματος Ευρωπαϊκού Εθελοντισμού Οπότε και σε αυτό θα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας για την επανεκκίνησή του, του προγράμματος αυτού του Ευρωπαϊκού Εθελοντισμού. Θα γίνουν διάφορα προγράμματα, πιλωτικά έργα σε όλη την Ευρώπη. Και εμεί δυστυχώ βέβαια δεν έγινε η Ευρωπαϊκή, το Ευρωπαϊκό Έτο Εθελοντισμού που θέλαμε εμεί και η Λευκή Βίβλο από την Κομισιόν. Αλλά ελπίζουμε φέτο με την 20η επέτειο να επανεκκινηθεί το όλο πρόγραμμα. Ευχαριστούμε που ήρθατε να μα δείτε και θα αναμένουμε τις ε, πιο αναλυτικέ πληροφορίε που σας ζητήσαμε που θα ήταν χρήσιμο να δώσουμε στους μα. Σα ευχαριστώ πολύ για την εξαιρετική σας δουλειά.